The meeting at four o'clock. Okay. Right, if, if people could sit down, we'll proceed. Καλό καθίστε. Vote on the... Για να συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες για τις οδηγίες για τις προοπτικές. We are voting. Right, could I see all those in... Could you sit down, still a few more members. Λοιπόν, έχουν καθίσει όλα τα μέλη. Me. Με ακούτε φαντάζομαι, το μικρόφωνο μου είναι εντάξει. Βέβαια μιλάνε πάρα πολύ και δεν διακρίνεται ορισμένοι από εσά καλά τη φωνή μου από ό,τι φαίνεται. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την οδηγία για τις προοπτικές. Θα ξεκινήσουμε με την F συμβιβαστική. Ποιοι είναι υπέρ F συμβιβαστική. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 94. Ποιοι είναι υπέρ της 94. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 16 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η συμβιβαστική G αγγλικά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 98 έχει αποσυρθεί. Οπότε πηγαίνουμε στην 99. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 102 αποσύρθηκε 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 103 και 104 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι γίνεται δεκτή αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 103 και 104. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Αντικαθιστώ κάποιον, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να ψηφίσω. Ψηφίζω για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν το ξέρω. Έτσι κι αλλιώς τέλειωσε η ψηφοφορία για τώρα. Σχόλια χωρίς μικρόφωνο στην Σοπάστε στο πάστε για να ελέγξουμε τους αριθμούς για να δούμε αν τυχόν ψηφίζει κάποιος που δεν πρέπει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τέλειωσε η ψηφοφορία, 25 υπέρ, 18 κατά. Δεν νομίζω ότι η ψήφο σα θα διαφοροποιούσε κάτι. Συνεπώς γίνεται δεκτή η διπλή αυτή τροπολογία. Περνάμε τώρα στην 105. Και είναι υπέρ. Κατά. αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 105. Τέλος της ψηφοφορίας. Είκοσι υπέρ, είκοσι κατά. Απορρίπτεται. 106 και 107 ταυτόσιμες ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109-110 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Συμβιβαστική H αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Περνάμε στην 117. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συγγνώμη, έχασα κάτι, πρέπει να πάω λίγο πίσω στη συμβιβαστική B αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα περνώ στην 118. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 124 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ της 22 κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική ή ε δηλαδή αγγλικά υπέρ κατά δεκτή 133 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 25 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 26 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 134 καταπίπτει. Ε, η 27 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική κάπα έχουμε μια προφορική τροπολογία από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι στο γραπτό κείμενο που έχετε μπροστά σας. Ο εισηγητής είναι κατά. Τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είμαι κατά. Απλά θα ψηφίσω κατά. Λοιπόν, δεν είστε κατά, θα ψηφίσετε κατά. Σας καταλάβαμε. Συμφωνείτε δηλαδή ε, με το να ψηφιστεί η προφορική τροπολογία. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε, το ελέγχουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία. Πέρα της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή η προφορική τροπολογία. Γίνεται πλέον δεκτή. Λοιπόν, το κάπα μαζί με την προφορική πλέον έγινε δεκτή. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε το κάπα με την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα πηγαίνουμε στην 150. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 153 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική γιώτα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα έχουμε μία πρόταση για ομαδική ψήφο από την 40 μέχρι την 67 έχει συμφωνηθεί να υπάρξει ομαδών ψηφοφορία από την 40 μέχρι 67 και είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή η ομάδα αυτή των τροπολογιών. Περνάμε τώρα στην 68. και είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Τώρα φτάνω στη συμβιβαστική α. Ποιοι είναι υπέρ τη συμβιβαστική α. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική γάμα C, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Οι 7 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 8 έχει αποσυρθεί. Η 76 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 78 και 79. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική J αγγλικά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλιστές νομίζω απέχουν, δεν ψηφίζουν. Α, είστε υπέρ. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβιβαστική J. Πέρα της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Απρόβλεπτη η ψηφοφορία. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεν ψηφίζει κανείς. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 85. Όχι. Για μια στιγμή. Ναι. 85. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 και 87 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 12 και 88 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική δέλτα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. 15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα θα γίνει ψηφοφορία για το σύνολο του τροπολογηθέντος κειμένου. που είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου όπως τροπολογήθηκε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 39 υπέρ 6 κατά. Και για το νομοθετικό ψήφισμα τώρα, πάλι ηλεκτρονικά. Ξεκινάμε. Πέραση της ψηφοφορίας. «38 υπέρ 6 κατά».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 We, we now have the vote. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα έχουμε την ε, ψηφοφορία για τη δική μου έκθεση. Για το διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και ίσως θα πρέπει να αναλάβει ο Αντιπρόεδρος τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Μπορούμε να ψηφίσουμε το κείμενο ολόκληρο, on block, πρόεδρε. Αν δεν έχετε αντίρρηση, ηλεκτρονικά. Καλώς λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για ολόκληρο το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Πρώτη εναλλακτική προσέγγιση. κατά αποχές Παράγραφος 2. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θετολογική σκέψη 1 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ετυλογικές σκύψεις ε, να... μέχρι 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία, 37 υπέρ, 3 κατά Οπότε τελειώνει η ψηφοφορία. Εδώ και δίνω και πάλι το λόγο στην κυρία Σάρων Μπόλς. Κύριε Κλίντς, Πρόεδρε, θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους της Επιτροπής μας ότι η Επιτροπή μας και δεν είναι η πρώτη φορά ε, με μεγάλη σοφία ψήφισε στα αισθητοτηρικές σκέψεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που όριζαν τα άρθρα στο διατακτικό. Δύο φορές επαναλαμβάνω. Δηλαδή έχουμε στην έκθεση ε, ασυνέπεια, εισαγάγει, λέμε κάτι στο αιτιολογικό που δεν υπάρχει μέσα στην, ε, στο διατακτικό και τούμπαλιν. Θα τα δούμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Ίσως πρέπει με τον τριμερή διάλογο να τα ρυθμίσουμε. Ήθελα πρώτα να προειδοποιήσω του συναδέλφου ότι διαπράξαμε μέγα σφάλμα. Έτσι λοιπόν έχετε και την ευκαιρία όπως σας βολεύει να τοποθετήσετε τη μία από εδώ και την άλλη από εκεί στον τριμερή λέει η πρόεδρος κυρία Βόρτμαν Κούλ. Κοιτάξτε, άλλο άρθρο, άλλο αιτιολογική σκέψη. Το άρθρο έχει σαφέστατη πλειοψηφία και νομίζω θα πρέπει να ε, υπερέχει της ε, αιτιολογικής σκέψης γεραρχικά. Καλώ, λέει ο Πρόεδρο. Αν έχετε την καλοσύνη, τώρα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη, που είναι η ανταλλαγή απόψεων για την επιτήρηση μια και έχουν παραταθεί οι προθεσμίε για την κατάθεση τροπολογιών και έχουμε και τόσες πολλές τροπολογίες, κινδυνεύουμε τώρα να μην έχουμε έτοιμη ε, την μετάφραση για τη δεύτερη εξέταση των τροπολογιών που έχει αρχικά προβλεφθεί, που βρίσκεται τώρα στο πρόγραμμά μας για τις 12 Απριλίου για το πακέτο για την επιτήρηση. Επομένως θα χρειαστεί να αναβάλουμε για την 22 Απριλίου, 5η στο Στρασβούργο. Ξέρω ότι δεν σας βολεύει πολύ η μέρα αυτή, πλην όμως ήταν η μόνη δυνατή ημερομηνία. Ως ε, μόνη εναλλακτική θα ήταν 3 και 4 Μαΐου, άλλη ημερομηνία που θα μπορούσα σας προσφέρω, αλλά θα έπρεπε να αναβληθεί αναλόγως και η ψηφοφορία στην Οικονομική Επιτροπή τον Ιού, για τον Ιούνιο και μετά θα πήγαινε στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο όλο αυτό το θέμα. Ενώ θέλουμε ή δυνατό να το κλείσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Επομένω, 22 Απριλίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στο Στρασβούργο. 22 Απριλίου. Αυτό λοιπόν αποφασίζεται. I think what we'll do is just go... Και νομίζω το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε μια ματιά στις εκθέσεις, στη σειρά που έχουν στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε πρώτα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών με εισηγητή τον Χωσέ, τον Αντιπρόεδρο. 10, 20, 30, 40, 50. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Τρεις παρατηρήσεις έχω καταρχήν να κάνω και μετά να αναφερθώ σε δέκα θέματα μέσα στα οποία θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όλες τις τροπολογίες. Οι παρατηρήσεις μου καταρχήν. Προσπαθούμε να δουλέψουμε γρήγορα ώστε υπό Ισπανική Προεδρία να εγκριθεί αυτό το εποπτικό πακέτο. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια δυσκολία. Η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώθηκε πριν αρχίσει να ισχύει η Λισαβόνα και πρέπει συνεπώς να προσαρμοστούμε τώρα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Στην προηγούμενη κατάσταση ίσχυε η επιτροπολογία, η διαδικασία λαμφαλούζη, ενώ τώρα έχουμε διαφορετικές νομικές καταγορίες, ιδιαίτερα ε, με πράξεις εφαρμογής. Η τρίτη μου παρατήρηση έχει να κάνει με το εξή. Όλοι οι ηγητές αποφασίσαμε ότι θα δουλέψουμε πάνω στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι πάνω στη συμφωνία του Συμβουλίου. Τώρα, πρώτη θεματική κατηγορία έχει να κάνει με το συστημικό χαρακτήρα του συνόλου των οργάνων που έχουν να κάνουν με την εποπτεία. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τις εθνικές αρχές, με το συστημικό κίνδυνο, τις τρεις επιτροπές, τη μεικτή επιτροπή και ό,τι έχει να κάνει με το πακέτο της εποπτείας. Και όλες αυτές τις τροπολογίες τις εξετάζω συνολικά γιατί είναι ένα πρώτο βήμα προς μια ενιαία εποπτεία που έχει προχωρήσει. Οπότε έχουμε τις τροπολογίες Skinner για την Μικτή Επιτροπή, ε, τις ε, τροπολογίες όσον αφορά για την, ε, τον ενίο χώρο και την τροπολογία της Αντιπρόεδρου που αναφέρεται στις έκτακτες διαδικασίες όταν πρόκειται για συστημικό κίνδυνο. Το πρώτο θέμα λοιπόν έχει να κάνει με τον Ευρωπαίο Ενίο Χώρο και έχουμε την, ε, τον κατακαιρματισμό των ρυθμίσεων που έχουμε σήμερα. Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές. Πρώτα απ' όλα, πρωταγωνιστική, πρωταγωνιστικό ρόλο στην ε, αρχή τραπεζών, που γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα. Ε, διαβουλεύσεις πριν καταλήξουμε σε τράπεζα και μελέτες αντικτύπου για να πω ότι επικοδομητικά αντιμετωπίζω την έκθεση Σκίνερ. Προτείνω τώρα, όταν η Επιτροπή πρέπει να επικυρώσει το Κοινοβούλιο θα αποτελεί, θα αναλαμβάνει ένα ρόλο ελεγκτικό. Και θα συνεργαζόμαστε με τον αρμόδιο επίτροπο και θα του ζητάμε να μας πει σε τι αποκλίνει και σε τι όχι. Εννοείται ότι και το Συμβούλιο μπορεί να κάνει ακριβώς το ίδιο. Το τρίτο μου σημείο είναι ότι για να αντισταθμίσουμε όλη αυτή την εξουσία που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Τραπεζών, θέλουμε να υπάρχει και έλεγχος των αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει να έρχεται εδώ λοιπόν ο ε, πρόεδρος και να έρχεται και να μας λέει τι έχει κάνει στην εντολή του. Όσον αφορά τώρα τις τεχνικές προδιαγραφές. Με τον ε, συνάδελφο και συμπατριώτη Μπρεσέδο υπάρχουν σημεία με τα οποία συμφωνούμε και σημεία με τα οποία διαφωνούμε. Οι τεχνικέ προδιαγραφέ αναφέρονται σε νομικέ πράξει, οι οποίε δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στρατηγική σημασία αποφάσει ή πολιτικέ αποφάσει που αυτέ τι παίρνουν τα δύο νομοθετικά σώματα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Με αυτό συμφωνούμε. Διαφωνούμε όμω το εξή. Εγώ βλέπω όλε τι τεχνικέ προδιαγραφέ, τι βλέπω σαν πράξει βάσει του άρθρου 290. Ο συνάδελφο Πρεσέδο τι χωρίζει σε δύο κατηγορίε. Εκείνε που αντιστοιχούν στο άρθρο 290 και εκείνες που, ε, που έχουν σχέση με το άρθρο 291 περισσότερο. Το πρόβλημα είναι τεχνικής φύσεως δηλαδή. Εδώ ζητάω η Γραμματεία των Νομικών Υπηρεσιών και της Δηματικής Επιτροπής να μας πούνε τελικά ποια θα ήταν η καλύτερη λύση σε αυτή την περίπτωση. Έρχομαι τώρα στους προσανατολισμούς και συνεχίζω εδώ με τις τροπολογίες των σοσιαλιστών που έκανε ο συνάδελφος Πρεσέδο. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε οι προσανατολισμοί να συμπεριλαμβάνουν τις πράξεις που δεν είναι κανονιστικές. Σκέφτομαι για παράδειγμα την, ε, τις αμοιβέ των εκτελεστικών οργάνων. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένας προσανατολισμός και όχι σύσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ώστε οι προσανατολισμοί αυτοί να είναι δεσμευτικοί τελικά. Υπάρχει ο πρόεδρος της αρχής ο οποίος θα μας πει τι προσανατολισμούς ε, επέλεξε και ε, σε ποιους δόθηκε συνέχεια και σε ποιους δεν δόθηκε συνέχεια. Η αμοιβή των ε, εκτελεστικών θέσεων, για παράδειγμα. Ατομικές αποφάσεις τώρα. Εδώ το πρόβλημά μου και τα προβλήματα που μου έθεσαν οι ομάδες έρχονται κυρίως από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές Άγγλους και έχουν να κάνουν με το θέμα των αποφάσεων που έχουν να κάνουν με ατομικές θεσμικές αρχές, εφόσον ο εθνικός επόπτης δεν έδωσε σημασία στις συστάσεις που έκανε ο εθνικός επόπτης. Στην περίπτωση που έχουμε κάτι τέτοιο, οι συστάσεις του επόπτη δεν πάνε στα σκουπίδια, πρέπει η αρχή τραπεζών να απευθυνθεί στο θεσμικό όργανο και να του ζητήσει να, εγκρί, να υιοθετήσει, να μην υιοθετήσει κάτι. Το αντεπιχείρημα βέβαια έχει να κάνει με τη νομική βάση. Αλλά είναι αδύναμο, διότι ούτε το Σεβούλιο, ούτε η Επιτροπή είπαν ότι θα υπάρχει νομική βάση όλες τις περιπτώσεις. Σε ορισμένε ναι, σε ορισμένε όχι. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη διάκριση βέβαια που γίνεται. Ίσως εκεί που υπάρχουν περισσότερα προβλήματα να έχει να κάνει με τη νομική βάση στην περίπτωση κοινοτική παράβαση. Και το επιχείρημα είναι ότι υπάρχει ήδη μια διαδικασία βάση του άρθρου 258, διαδικασία κυρώσεων. Η διαδικασία σε εθνικό επίπεδο είναι σίγουρα πάρα πολύ αργή και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσει του χρηματοπιστωτικού κόσμου σήμερα. Γι' αυτό και υποστηρίζω εγώ αυτό που υποστηρίζω. Δεν είναι θέμα νομικής βάσης, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Έρχομαι τώρα στην εποπτεία, αλλά όπως έχω ξαναπεί, η έκθεση ήταν Έρχομαι στο Βρετανικό, δηλαδή μετά το παράδειγμα της Λέμαν που είχαμε, που η πτώση της ε, οφείλεται στα γεγονότα στο Λονδίνο. Εδώ δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Ή που στην αφιτρίωνα χώρα δίνουμε περισσότερες αρμοδιότητες για τον έλεγχο ή ενισχύουμε το ρόλο των συλλογικών αρχών εποπτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή λύση, κατά τη γνώμη μου, αντιστοιχεί με αυτό που από το 2000 λέμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι επήγη. Επήγη σήμερα όσο ποτέ. Και δεν θέλω εδώ να σας πω ότι εγώ έλεγα το 2000, θα σας πω ότι έλεγε ο Μάρκοβαν που είναι σκιώδης για εκ μέρους των ε, σοσιαλιστών που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν όλα κινούνται τόσο πολύ γρήγορα, εμείς θα πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι συμφωνούμε η αρχή τραπεζών να έχει μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι είχαν μέχρι τώρα οι εθνικές εποπτικές αρχές και να έχει τη δυνατότητα διαμεσολάβησης με δεσμευτικό χαρακτήρα και να μπορεί δηλαδή να παίρνει αποφάσεις τέτοιες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή. Ποια είναι η πρόταση. Η πρόταση είναι ότι εκεί όπου υπάρχει συστημικός κίνδυνος, εκεί όπου μπορεί να καταρρεύσει τελικά το σύστημα, αυτοί οι οργανισμοί βρίσκονται υπό την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, η οποία μέσω των εθνικών εποπτών, για να μην υπάρχει περιττή γραφειοκρατία, θα δρά στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα αποφασίζει ακριβώς ποιοι θα κάνουν τι βάσει των κριτηρίων που καθορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από οποιοδήποτε άλλο που έχει αρμοδιότητα για να καθορίζει ποιες θα είναι οι αρμόδιες αρχές. Γιατί τώρα έχουμε Ευρωπαϊκή Αρχή. Για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι οι τράπεζες που οδηγούν σε συστημικούς κινδύνους είναι διαφορετικές. Δεύτερον, γιατί είναι αναγκαίο να μην έχουμε από τη μια μεριά οργανισμούς που δρούν μέσα σε ένα χώρο χωρίς σύνορα και άλλες όπου δρούν με εθνικά σύνορα. Και τρίτον, επειδή έχουμε την ελληνική περίπτωση και ορισμένες τράπεζες και η ελληνική τράπεζα μπορεί να μαγειρεύει τα δημοσιονομικά, οπότε αυτό θα γινόταν πολύ πιο δύσκολα εάν υπήρχε η εποπτεία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο εθνική εποπτεία. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν έχουμε καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα. Και γι' αυτό και θέλουμε να έρθει και κάποιος να εξηγήσει. Τώρα, Έρχομαι στο ταμείο, το οποίο θα βοηθήσει να πληρώνονται χρήματα σε περίπτωση κατάρρευσης ορισμένων χρηματοδοτικών ε, ιδρυμάτων. Τα χρήματα θα είναι από τις τράπεζες. Οι τράπεζες θα πληρώνουν έτσι κι τα χρέη αυτού του ταμείου. Πάντως την πρόταση αυτή θέλω εγώ να την επεκτείνω και στην περίπτωση των ασφαλίσεων που εξετάζει η έκθεση Σκίνερ. Τώρα τι γίνεται με το Συμβούλιο. Με το Συμβούλιο πάμε καλύτερα από ό,τι πηγαίναμε. Το Συμβούλιο βρισκόταν πολύ μακριά από τις δικές μας θέσεις, αλλά τελικά ενέκρινε πριν από μερικές μέρες τη στρατηγική 2020, που στο σημείο 4.2 λέει ότι για να βελτιωθεί η διαχείριση των οικονομικών κρίσεων και λαμβάνοντας ε, υπόψη τον τομέα πρέπει να βρεθούν οι σωστές λύσεις από τον ίδιο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Από εκεί θα χρηματοδοτηθεί το Ταμείο λοιπόν. Τέλος, οι διεθνείς σχέσεις νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι για το ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει με μία φωνή. Αλλιώς κινδυνεύουμε να πρέπει να χορέψουμε στη μουσική που παίζουν άλλοι. Τέλος, κυρία Πρόεδρε. Είδατε ότι περιορίστηκα, αλλά θέλω να προσθέσω ένα πράγμα. Την συμμετοχή στην εποπτεία. Η έκθεση που μας έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο επικεντρώνεται πολύ στις τράπεζες. Όμως μην ξεχνάμε ότι προορίζονται τα χρήματα κυρίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επίσης να συμμετέχουν στην ομάδα συμφερόντων και να ακούγονται και αυτοί στα επιπληκτικά όργανα για να μπορούν και αυτοί να έχουν λόγο για το κόστος ε, το πιστοτικό. Τώρα ξεκινάει η πραγματική δουλειά, κυρίες και κύριοι. Τώρα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις που θα είναι δύσκολες, διαπραγματεύσεις τις οποίες θα πάω με τις ιδέες τις οποίες περιλαμβάνει η έκθεσή μου και που πιστεύω ότι είναι σημαντικές, γιατί αλλιώς φυσικά δεν θα τις είχα βάλει στην έκθεσή μου. Από εδώ και πέρα είμαι στη διάθεσή σας για διάλογο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στον εισηγητή για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Σβέν. Καταρχάς, και προκαταβολικά θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και συνάφη μεταξύ της δουλειά που κάναμε όλοι οι συγητές εδώ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να αποφύγω τα όσα ε, ήδη έχουν καλυφθεί για να κερδίσουμε και χρόνο. Σε ένα σημείο θα ήθελα ιδιαίτερα να ε, ε, επιμείνω που έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί άλλαξε και με τις νέες τροπολογίες ότι Θέλουμε να ενισχύσουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, στο πλαίσιο των, ε, της stakeholder group ε, για να υπάρχει η σαφής παρουσία τους και να εξασφαλιστεί η ισότητα των συσχετισμών δυνάμεων εδώ. Μια ισορροπία στους σχετισμούς δυνάμεων. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, θεωρώ πολύ σημαντικό, εάν δούμε ιδιαίτερως ε, πόσο περιορισμένους ισχνούς πολλές φορές πόρους έχουν οι οργανώσεις για την προστασία των καταναλωτών και των δικαιώματων τους και αν αυτό το συγκρίνουμε με τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών. Έτσι λοιπόν η ανισότητα των ε, όπλων σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να παρέμβουμε για το δικό μας φυσικά συμφέρον έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η ισότητα. Η ιδιαίτερα στην Επιτροπή αυτή, στην Εποπτική Αρχή, ώστε να υπάρχει ε, ικανοποιητική εκπροσώπηση. Επίσης, θα θέλαμε να προσδιοριστεί ο τομέας επακριβώς, τον οποίο θα παρακολουθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων της και για να το πω στα αγγλικά, τα δικαιώματα των μετόχων, η, ε, εταιρική διακυβέρνηση, δημοσιονομικός, ε, παραλογιστικός έλεγχος, ζητήματα καθαρίσεων, ρυθμίσεων, ε, του short selling των παραγόγων και μια σειρά από πρότυπα που θα πρέπει να εισαχθούν στους ανωτέρω τομείς. Τρίτον, προτείνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάλι Στη συνεννόηση με τους ε, ενδιαφερομένους φορείς, να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μητρό, όπως προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες, στο οποίο και οι ε, παράγοντες της αγοράς θα μπορούν να βλέπουν ξεκάθαρα, θα ισχύει για όλη την Ευρώπη, εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει τιμωρηθεί, έχει υποστεί ποινική κύρωση για λόγους ε, πλημελούς συμπεριφοράς εάν υπάρχουν ζητήματα κατάχρησης ε, της κυριαρχής ε, θέσης στην αγορά, στις πόσες θέσεις και ούτω καθεξής. Επίσης, ε, στο θέμα του κατά πόσο θα πρέπει να απαγορευθούν κάποια προϊόντα χρηματοπιστωτικά, ύστερα και από τα όσα συστήσαμε σήμερα το πρωί, θα ήθελα να πω ότι δεν κοιτάμε να απαγορεύσουμε ή μάλλον να, επιβάλλουμε υποχρεωτική προεξαγγελία και πρώτερη έγκριση κάθε δυνατού προϊόντος που ενδεχομένως να ε, ε, μπαίνει στην αγορά. Όχι, αλλά εάν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, εάν δούμε ότι κάτι συμβαίνει στραβό και παράτυπο, θα πρέπει να είμαστε θέση να απαγορεύουμε την ε, ε, ε πώληση ενός διάθεσης του προϊόντος. Και θέλουμε, στο επόμενο σημείο, τα δικαιώματα των εθνικών αρχών εποπτείας να είναι αντίστοιχα με αυτά της Ευρωπαϊκής Αρχής. Δηλαδή θέλει, θέλουμε και η Ευρωπαϊκή Αρχή να έχει αντίστοιχα ε, δικαιώματα και ε, αρμοδιότητες. Να μπορεί να παρακολουθεί κάθε λειτουργία της αγοράς ώστε να αποφεύγει εσφαλμένες πρακτικές και να επιβάλλει υψηλές προδιαγραφές για όλους τους ε, παράγοντες της αγοράς, όταν αυτές δεν υπάρχουν. Άλλο σημείο, την απόφαση για την απόψή μας για το πρώτο, για το πότε υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν θα πρέπει να το αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το σύστημα, το Συμβούλιο μάλλον για τη διαχείριση των ε, κινδύνων. Και στο άρθρο 10 η νομοθεσία του άρθρου 1 παράγραφος 2 θα πρέπει να ε, την έχουν τα κράτη-μέλη όπως άλλωστε και τους όρους του ίδιου του κανονισμού. Επίσης στη συνέχεια ζητήματα εκπροσώπησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετοχής τρίτων κρατών για να συμφωνήσουμε με τα όσα είπε και ο κ. Μαρκάγιο νωρίτερα. Προχωρώ επίσης για να πω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες προδιαγραφές επιτήρησης ε, τρίτων κρατών και εφόσον αυτές προβλέπονται θα υπάρχει δυνατότητα της εκχώρησης του πλήρου εξουσίου δηλαδή. Επίσης η ομάδα των ε, εμπλεκομένων φορέων, των stakeholders ε, θα λαμβάνει τις απαιτούμενες αποφάσεις, θα έχει τακτικές συνεδριάσεις, υπάρχει μια διασφαιριστική δικλίδα με το άρθρο 23 όπου θα επαληθεύεται ότι ένα κράτος μέλος ε, εάν ένα κράτος μέλος έχει άμεση ή έμεση εμπλοκή μέσω της συμπεριφορά του ε, της δημοσιονομικής. Μετά θα έχουμε μια διαδικασία αξιολόγησης και ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη της αρχής όπου θα πρέπει βεβαίως να συστήσουμε με μεγάλη σοβαρότητα και το ζήτημα του ε, οπλοστασίου που θα προσφέρουμε σε αυτή την Επιτροπή, σε αυτήν την αρχή επιτήρησης. Η κοινή Επιτροπή και η ομάδα των stakeholder θα πρέπει να είναι σε θέση να καταθέτει προτάσεις και αυτά όλα τα βλέπετε σε μια αξιολόγηση που έχουμε στην έκθεση μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αναρωτιέστε τι θα κάνω. Θα ακούσουμε πρώτα τους εισηγητές και μετά θα περάσουμε στους σκιώδεις εισηγητές και στους τα υπόλοιπα μέλη. Αυτό είναι ένα πακέτο έτσι ώστε να ξέρουμε από την αρχή ποιοι θα μιλήσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από την αρχή εποπτείας συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Το πρώτο θέμα είναι το πόσο φιλόδοξοι είμαστε και τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο και να βρεθεί σε θέση ε, διαπραγμάτευσης όταν συναντηθούμε με το Συμβουλίο με μια κάποια δύναμη. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση, αν όχι να παίξουμε άμεσα τα χαρτιά μας, αλλά να προσπαθήσουμε να πείσουμε το Συμβούλιο να κάνει υποχωρήσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πραγματικότητα την οποία θα επιλέξουμε να κινηθούμε. Οι συνάδελφοι έχουν συμφωνήσει σε πολλά θέματα, αλλά υπάρχει ένα θέμα φιλοδοξίας θα έλεγα, δηλαδή ευρύτητας πεδίου αναφοράς και χρόνου. Επανέρχομαι στις παλαιότερες συζητήσεις που είχαμε για το κατεπήγον του να υπάρξει αυτή η αίθουσα, η έκθεση συγγνώμη, πριν το καλοκαίρι έτσι ώστε την 1η Ιανουαρίου του 2011 να έχουμε στη διάθεσή μας κάτι το συγκεκριμένο. Εγώ προέβλεψα ένα συγκεκριμένο, θα έλεγα, χρονισμό, σύμφωνα με τη δυνατότητα την οποία έχουμε, να φτιάξουμε μια πλατφόρμα στα πλαίσια της οποίας να κινηθούμε και είμαι φιλόδοξος αρκετά ότι θα μπορέσουμε την 1η Ιανουαρίου 2011 να έχουμε κάποια πρώτα πράγματα στη διάθεσή μας. Να έχουμε μια διαδικασία δηλαδή με έναν υπεύθυνο για τη διαδικασία αυτή, με μια δυνατότητα ταμιακής παρέμβασης. Θα δούμε αν θα το πετύχουμε. Έχω κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε και να φτιάξουμε κάτι το οποίο να έχει νόημα στις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο. Καταρχάς, ο πρόεδρος αυτού του, αυτής της εποπτικής αρχής θα πρέπει να επιλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει στα πλαίσια της ψηφοφορίας να ληφθούν υπόψη όχι μόνο κάποια τεχνικά επίπεδα, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε στενότερες σχέσεις ανάμεσα στις εποπτικές αρχές και οι εποπτικές αρχές ε, πολλές φορές ε, εξαρτώνται από το να καταψηφίζουν η μία την άλλη, ενώ η πραγματικότητα είναι η αναζήτηση της ομοιοτυπίας και της συμβατότητας. Μετά, να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε σωστά τις ομάδες των εμπλεκομένων, των stakeholders. και θα πρέπει να υπάρχει επίσης και μια, μια έκθεση μειοψηφία ή εκθέσεις μειοψηφία από τις ομάδες των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων. Για το 12α υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ μας. Έχω κάνει μια συμβιβαστική πρόταση την οποία συνυπέγραψε και ο συνάδελφός μου και ο Σπεσέρα από την δική μου πολιτική ομάδα. Further, in terms of... Ο κύριος Πεσέδο έτσι ώστε να υπάρχει μια ρήτρα ε, που μας δίνει τη δυνατότητα μέσα σε τρία χρόνια να αναθεωρήσουμε την πρόταση, να καταστήσουμε τη διαδικασία αυτή ολοκλήρωσης ε, πιο ισχυρή και να καταλήξουμε ίσως και σε μία εποπτική αρχή. Αυτό πρέπει κάποτε να γίνει, δεν μπορεί να γίνει άμεσα, πρέπει να γίνει σταδιακά. Η τροπολογία λοιπόν μας επιτρέπει και να έχουμε όραμα και να έχουμε φιλοδοξίες και να είμαστε ρεαλιστές. Πολλοί θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου με αυτό. Δεν ξέρω τι πλούτος υπάρχει σχετικά με την συνταξιοδιωτική βιομηχανία, αλλά πολλοί μιλάνε για 55-3 ευρώ στον τομέα των ασφαλιστικό. Καταλαβαίνετε δηλαδή με τι ακριβώς ποσά έχουμε να κάνουμε όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα ταμείο. Πολλοί διαφωνούν με αυτά που λέω, αλλά νομίζω ότι εγώ βλέπω κάποια γεγονότα. Τώρα για κάποιες ίσονες τροπολογίες. Θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις εις βάρος συγκεκριμένων οργάνων και θεσμών για μη εφαρμογή κοινοτικών κανόνων. Αυτό θα αφορά πιστοτικά ιδρύματα, οικονομικά ιδρύματα ιδιαίτερα στις χώρες μέλη που δεν σέβονται τους κοινωνικούς κανόνες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στα σώματα τα οποία ήδη λειτουργούν σήμερα. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να συνεχίσουν να παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του διακανονιστικού πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει να γίνονται σωστοί έλεγχοι και εποπτείες αποφάσεις για ισοτιμίες και γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν λοιπόν στο επιθυμητό επίπεδο όλες αυτές οι αποφάσεις και τα όργανα αυτά να παίξουν τον ρόλο που παίζει το ΣΥΟΠΣ σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπλέκεται στο ΣΥΟΠΣ και θα πρέπει να εμπλακεί ακόμα περισσότερο και στη δημιουργία της εποπτικής αρχής. Δεν γίνεται αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα και θα ήθελα να εμπλακούν ακόμα βαθύτερα. Όλες οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί για όλες αυτές τις εποπτικές αρχές. και αφορούν την μεικτή συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί. Υπάρχει μια κάποια συνένεση. Έχουμε κάποιες δυνατότητες να συμφωνήσουμε σε επίπεδο νομικών μέσων και να δημιουργήσουμε την διαδικασία η οποία θα μπορέσει να σκληρύνει και να ολοκληρώσει την εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς ε, να εφεύρουμε θα έλεγα έναν επόπτη Ευρωπαίο ε, από τη μία μέρα στην άλλη κάτι το οποίο δεν θα ήταν ρεαλιστικό. Ευχαριστώ. Όντως χρειάζεται η μακροσυστημική επιτήρηση. Σόφη. Ναι, η συζητήσεις τώρα για το δικό μας θέμα της μακροπολιτικής εποπτείας του πρωτοπροστατικού συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε κάποια σημεία ενδεχομένω όπου μπορεί ο καθένας να δίνει την έμφαση σε άλλο σημείο. περιορισμένα όμως σημεία διαφοραοποίησης. Στην έκθεση Λαροζιέρα έγινε μια πρόταση, την οποία ακολούθησε και η Επιτροπή και δεν αμφισβητεί πιστεύω κανείς, δηλαδή ότι η μικροοικονομική επιτήρηση τίθεται υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας με σημαντικό ρόλο και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, κυρίως λόγω της ε, ευχέρειας που έχουν να είναι ο τελευταίος ε, διεξόδουδαν στις... Δηλαδή πρέπει κανείς να γνωρίζει τι θα κάνει σε περίπτωση κρίσης, αν θα απευθυνθεί στην τράπεζα ή μη. Ε, εγώ ήθελα να δώσω κάποιες συγκεκριμένες, ε, κάποια συγκεκριμένη έμφαση ως προς τον κεντρικό τραπεζίτη, την κεντρική τράπεζα δηλαδή. Αυτή είναι η βάση με την οποία εργαστήκαμε και πάνω στην οποία θα θέλαμε ίσως περιορισμό, θα θέλαν ορισμένοι ίσως περιορισμό της ε, επιρροής. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε, να αναζητήσουμε μια ισορροπία αφενός μεταξύ της ανάγκης για περισσότερη διαφάνεια, γιατί υπάρχει ανάγκη ε, για διαφύλαξη και της, του απορρίτου ορισμένων ε, πληροφοριών αλλά και της ανεξαρτησίας. Ταυτόχρονα εγώ δεν θα ήθελα να εισαγάγω ε, ως ίσους μέσα στα όργανα αυτά εκπροσώπους του βιομηχανικού τομέα, της οικονομίας κτλ. Αλλά ίσως κάποια άτομα θα μπορούσαν να διαφυλάξουν μια ε, ένα κάποιο άνοιγμα πνεύματος, ίσως θα έπρεπε να δούμε από εκεί ε, σε εάν οι θέση του θα είναι μέσα στο Γενικό Συμβούλιο ή στην Διευθυντική Επιτροπή. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι πάλι ζήτημα διαφάνεια, ε, το αν θα αρκεστούμε σε ένα ιστορικό ε, συμβουλευτικό όργανο το οποίο θα παρτίζεται λίγο πολύ από το σύνολο των εμπειριών των 27 ε, κεντρικών τραπεζών ή αν θα ε, ζητούμε και την εξωτερική πραγματογνωμοσύνη από τους ε, πανεπιστημιακούς. Έχοντας ακούσει ο Μάριο Ντράγκη και τον, Μίστη του Καν, όπως όλοι σας βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ καταλήγω ότι επιβεβαιώνεται η αρχική μου πρόταση για πανεπιστημιακούς πανεπιστημιακούς καθηγητές του, του ε, παγκοσμίου κύρους και βλέπουμε εντύπωση ότι και οι δύο αυτοί ομιλητέ, ο οποίο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, λένε ότι πρέπει να αναπτύξουμε νέους, νέα οράματα για την επιτήρηση. Τρίτο θέμα. Λαμβάνεται τώρα η απόφαση για την ε, ε εποπτεία ή ξεκινούμε από τα δεδομένα που έχουμε ήδη. Η έκθεση Λαροζιέρ μιλάει μάλλον για την διατήρηση των τριών επιτροπών Λαμφαλούς, την ενίσχυσή τους των αρμοδιοτήτων και των, ε, ε του αρχιτεκτονήματός τους, αλλά από την άλλη λέει ότι συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Εγώ νομίζω ότι έτσι ε, περιορίζουμε πολύ τις δυνατότητές μας, γιατί όταν έχουμε τρία διαφορετικά όργανα κατεστημένα σε διαφορετικές πόλεις, τι να τους πούμε ότι πρέπει να επεκταθούν, να αναπτύξουν δραστηριότητες κτλ. Για να έρθουμε τρία χρόνια αργότερα με την αναθεώρηση να τους πούμε «Α, τελικά όχι, πρέπει να συνεργάζεστε περισσότερο». Δεν έχει νόημα όλο αυτό και νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο οι επιλογές θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτέ, περισσότερες ε, μπροστά μας. Ο αντιπρόεδρος που ψήφισε ο αντιπρόεδρος σήμερα το πρωί μας μίλησε για τη δυνατότητα ενός Twin Peaks, μιας ε, διπλής αιχμής θα σήμαινε δηλαδή αυτό δύο, όχι τρία βέβαια όργανα, αλλά πάντως έβλεπε μια τέτοια λύση. Ε, χωρίς να έχουν κλείσει όλα τα θέματα, νομίζω ότι μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση που δεν θα μας κλείνει για το μέλλον τις επιλογές. Ευχαριστώ τους αδέλφους που κατέθεσαν τις σχετικές προτάσεις. Ε, βλέπω ότι υπάρχει μια δυνατότητα η Επιτροπή για, το Συστημικό Κίνδυνο από την αιγίδα της ε, Γενικής Τράπεζας που βρίσκεται στη Φραγκφούρτη και νομίζω ότι θα ήταν λογικό να επιλέξουμε κάτι που είναι σημαντικό βέβαια για τον πολίτη, μια λογική περισσότερο της αποτελεσματικότητας και όχι της αναγνώρισης του κύρους της μίας ή της άλλης πρωτεύουσα ε, κράτους. Επίσης, για τους ε, εισηγητές που είναι υπεύθυνοι για τις επιτροπές μικροεποπτείας, ε, και το, πώς ορίζεται το κατεπήγον που αναφέρθηκε νωρίτερα. Μα η, Επιτροπή, η έκθεση πάνω της Επιτροπής για το Συστημικό Κίνδυνο πρόβλεπε ήδη την ε, δυνατότητα ταξινόμησης κινδύνου, δηλαδή να λέει αν υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος ότι είναι, να τον περιγράφει σοβαρό, να κάνει το χαρακτηρισμό δηλαδή του κατεπήγοντος. Ε, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το πράξει και μάλιστα σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια όργανα και τις αρχές και όχι κατά αποκλειστικότητα. Αυτά. Κατά τα άλλα θα δούμε και άλλες ε, φορές τους σκιώδεις. Περιμένω κάθε πρόταση να την ακούσω να τη συζητήσω. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά που βλέπουμε με την κερδοσκοπία εις βάρος του ευρώ, εις βάρος ενός κράτους μέλους, εάν τυχόν υπάρχει όπως να επαναληφθούν και στο μέλλον, όπως άλλωστε εκφράστηκε χθε ο φόβος, ε, που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την ε, σταθερότητα, για τη στερεότητα ενός κράτους ολόκληρου, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κανείς δεν έχει την απόλυτη αλήθεια στη διάθεσή του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλά μπορούμε να δούμε σαν παραδείγματα, αλλά πάντως πρέπει να επιλέξουμε τις λύσεις εκείνες οι οποίες θα αποτρέψουν στο μέλλον τέτοιου τύπου δυσάρεστες εξελίξεις. Ευχαριστώ. Um, thank you very much. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στα ειδικά καθήκοντα της Κεντρικής Τράπεζας, ε, τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ο κύριος Τρεμόσα είναι ο εισηγητής, αλλά είναι σκιώθης και για άλλα θέματα. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου δύο λεπτά να σας απασχολήσω. Η έκθεσή μου είναι ένα σύντομο σχέδιο έκθεσης ουσιαστικά. Είναι για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διάφορα ειδικά καθήκοντα όσον αφορά την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου προβλέπεται μια στενή σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Εμείς μάλιστα προτείνουμε πρόεδρος του Συμβουλίου αυτού να είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν συναδέλφου ευρωβουλευτές που με βοήθησαν προσφέροντας μου κείμενα άρθρα οικονομικά για να μου πούν ότι υπάρχει ασύμβατο ανάμεσα στη σταθερότητα τιμών και την οικονομική σταθερότητα. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο αυτό έχει σαν στόχο να διατηρήσει σταθερές τις τιμές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συγγνώμη. Ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έχει σαν στόχο να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Είναι ασύμβατα, μου είπαν αυτά τα δύο. Ίσως όσο δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση, κάτι που να τις μοιάζει, πιστεύω και εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι το μόνο ανεξάρτητο όργανο σήμερα που να έχει την ε, ηθική ικανότητα να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην μελλοντική ευρωπαϊκή εποπτεία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όπως είπα και πριν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέρφους που με βοήθησαν να δω ότι υπάρχει αυτό το ε, ασυμβίβαστο. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώς γι' αυτό προτείνω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει αυτό το σημαντικό ρόλο ως μοναδικός οργανισμός που να έχει την δυνατότητα να εποπτεύσει. Προτείνω μια τροπολογία στην ίδια μου την έκθεση, με την οποία προτείνω ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου να έρχεται κάθε εξάμεινο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσει για την οικονομική εποπτεία. Πέρα δηλαδή από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που όπως έρχεται τώρα θα συνεχίσει να έρχεται κάθε τόσο. Κατά τη γνώμη μου, και συμφωνώ με αυτά που είπε ο Στράσκο την προηγούμενη εβδομάδα, στην Επιτροπή μας που είπε ότι η οικονομική εποπτεία είναι πιο σημαντική από την οικονομική ρύθμιση. Δεν έχει νόημα να έχουμε την καλύτερη δυνατόν οικονομική ρύθμιση χωρίς να έχουμε αποτελεσματικό έλεγχο και εποπτεία. Γι' αυτό εμένα με απασχολεί το εξή. Σήμερα το πρωί ο κύριος Κωνστάντσιο μας υπενθύμησε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν δίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, καθήκοντα εποπτικά. Δεν αναθέτει τέτοια καθήκοντα εποπτείας. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η εποπτεία να είναι ισχυρή, γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία να το πετύχουμε αυτό. Σε 5 σε 10 χρόνια, αν έχουμε άλλη οικονομική κρίση, σαν και αυτή που έχουμε σήμερα, οι κυβερνήσεις δεν θα έχουν περιθώριο για να βοηθήσουν. Δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία για να διορθώσουμε τη ζημιά από μια κρίση σαν και αυτή που έχουμε σήμερα τέτοιου μεγέθους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Now we move on to... Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στις εξουσίες των εποπτικών αρχών αυτών και τροπολογίες σε μία σειρά οδηγιών, το Omnibus 1. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε σχέση με το Omnibus, ναι. Για τα άλλα θα σας πω μετά. Το Omnibus τι προσπαθεί να κάνει. Με 11 οδηγίες επιμέρους θέλει να συμπεριλάβει τόσο έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις των νέων αρχών. Είναι 11 τομαϊκές οδηγίες που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες και με τις αξίες. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για την ύπαρξη αυτών των αρχών, για τον συντονιστικό ρόλο που πρέπει να αναλάβουν οι αρχές αυτές, τη συνεργασία τους με τις ήδη υπάρχουσες ε, αρχές που προβλέπονται από τις τομαϊκές οδηγίες, τη διαμεσολάβηση για θέματα που έχουν να κάνουν με προσανατολισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και κυρίως να δούνε τους τεχνικούς κανόνες. Οι τεχνικοί κανόνες είναι εκεί που πρέπει να υπάρξει προσαρμογή, ανανέωση. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Μαργάγιο, οι προτάσεις ξεκίνησαν πριν να αρχίσει να ισχύει η Λισαβόνα. Και με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε δύο κατηγορίες τώρα. Έχουμε πράξεις που δεν υπήρχαν πριν. Ακριβώς επειδή είχαμε την αρχιτεκτονική λαμφαμουσή, ήταν επιτροπολογία που ρύθμιζε πολλά πράγματα με μία κατηγορία. Ενώ τώρα έχουμε δύο. Γι' αυτό λοιπόν αλλάζουν τα πράγματα και γι' αυτό και έχουμε σήμερα τις νέες αυτές πράξεις. Πριν είχαμε ρυθμιστικά, εφαρμοστικά μέτρα Πώς τώρα όλο αυτό το σύστημα συνδυάζεται με την οδηγία Omnibus. Η οδηγία Omnibus, παρόλο που ανταλαμβανόμαστε τα τέσσερα επίπεδα τη λαφαλουσή, μας ενδιαφέρει κυρίως το επίπεδο 2 και το 4, το 2 που είναι το ρυθμιστικό επίπεδο, κάτω από την νομοθεσία δηλαδή, και το 3 που πριν ήταν κατακαιρματισμένο σε διάφορες εθνικές αρχές που συνεργαζόντουσαν σε επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 από εδώ και πέρα θα είναι ένα επίπεδο δεσμευτικό και πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχουν οι τεχνικοί κανόνες και στο επίπεδο 2. Αυτό προσπαθήσαμε να λύσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στους τεχνικούς κανόνες. Καθορίσαμε λοιπόν κάποια κριτήρια με Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές. Μπορούμε πάντα να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις εφόσον τηρηθούν κριτήρια χρήσιμα για το μέλλον. Τα κριτήρια λοιπόν που έχουν καθοριστεί για να δούμε τους τεχνικούς κανόνες είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, όταν ένας τεχνικός κανόνας εξελίσσεται, είδαμε στις οδηγίες ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα νομοθετικής εξέλιξης. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Ένα επίπεδο που να είναι το τέος 2 και ένα επίπεδο 3. Γιατί στην εξέλιξη βλέπουμε ότι υπάρχουν επικαλύψεις. Δεν θέλουμε να τα βάλουμε όλα στην ίδια κατηγορία. δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μακρές διαδικασίες. Οπότε το βασικό, οι τεχνικοί κανόνες λειτουργούν στο επίπεδο 2 και 3. Στο επίπεδο 2 πρόκειται για ε, στάνταρ περιπτώσεις και το κριτήριο που χρησιμοποίησαμε είναι ότι οι πράξεις που ανατίθενται πρέπει να βασίζεται σε, ένα, σε κοινούς κανόνες, single Book. Πρώτον, να υπάρχουν οι ορισμοί. Οι ορισμοί να είναι συγκεκριμένοι και κοινοί. Δεύτερον, να καλύπτονται τα reporting και disclosure που να είναι κοινά. Η πληροφορία που πηγαίνει σε άλλους φορείς ή στις αρχές θα πρέπει να είναι η ίδια. ώστε η εποπτεία να γίνεται ομοιόμορφα. Και τρίτον, αυτή η κοινή και συνεπής εποπτική προσέγγιση πρέπει να φτάνει σε όλες τις αρχές που συμμετέχουν στο οικονομικό σύστημα για να μπορούν να συνεργάζονται. Αυτό είναι αναγκαίο για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Και από εκεί και πέρα. Αυτό είναι το single rule book, έτσι. Γιατί συνάδει μάλιστα και με το άρθρο 291 της συνθήκης, που λέει ότι υπάρχει συμπλήρωση με τις πράξεις που ανατίθενται των ήδη υπαρχόντων. Στο επίπεδο 3 λοιπόν θα αφήσουμε τις εφαρμοστικές πράξεις. Για αυτές τις δύο περιπτώσεις τεχνικών κανόνων, οι αρχές καθορίζουν προδιαγραφές σε επίπεδο 3 που είναι για την εποπτεία. Κάτι όμως το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε να οδηγεί σε συνοχή όλες τις πράξεις τις ρυθμιστικές. Αυτό που δεν έχω κάνει, γιατί ναι με για τα κριτήρια στην πρόταση της Επιτροπής, αυτό που δεν έκανα είναι να συμπεριλάβω κριτήρια που ήθελε η Επιτροπή μας. Γι' αυτό και υπάρχει η σχετική τροπολογία, η οποία ξεκινάει από το κεκτημένο το οποίο έχουμε σήμερα στις διαδικασίες, που είναι η έγκαιρη παρέμβαση, Και έτσι έχουμε αυτές τις τροπολογίες. Για την οδηγία Omnibus λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες για να πετύχουμε συμβιβασμούς. Η Νομική Επιτροπή θα έχει επίσης τροπολογίες, ένα πακέτο από ό,τι φαίνεται, σημαντικό, με στόχο να οδηγήσει σε συνοχή τις τροπολογίες της Νομικής Επιτροπής, τις δικές μας και να καταλήξουμε έτσι σε μια λύση με τους εισηγητές που έχουν αναλάβει τις κύριες εκθέσεις. Um, oh, uh, Καλώς λοιπόν, βλέπω στον κατάλογο μου και έχει ζητήσει το λόγο η Βίκη Φόρντ. Sorry about that. The, um, you get fit running around the Parliament in between two different. <laughs> Αναγκάζομαι να παρακολουθώ δύο διαφορετικές επιτροπές. Συγγνώμη που έλειπα. Να σταθώ λίγο σε τροπολογίες τις οποίες δεν έχω ακόμα δει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα τεράστιο πακέτο. «1527». Οπότε προς το παρόν νικά ο Ζωαπόλου. έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία όλες αυτές οι τροπολογίες και γι' αυτό υπάρχει και αρκετή συνένεση θα έλεγα σχετικά με τη συνεργασία των ελεγκτικών αυτών αρχών και είναι σημαντικό να υπάρχει αρκετή συνένεση γύρω από τα θέματα αυτά. Είναι τόσο σημαντικό λοιπόν που θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν, στην πρώτη ανάγνωση θα λέγαμε. και οι περισσότερες τροπολογίες τις οποίες έχω καταθέσει μας ε, φέρνουν πιο κοντά στις θέσεις του Συμβουλίου για να ξεκινήσει η διαδικασία. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε εμά που πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή θα είναι εξελικτική και σε κάποιους που θέλουν να υπάρχουν ρήξεις. Και άκουσα αυτό που είπατε και για την ρήτρα αναθεώρησης μετά από λίγα χρόνια. Εμείς δεν πήραμε φυσικά το κείμενο του ε, Συμβουλίου και υποβάλαμε εκ νέου κάθε τροπολογία που είχαμε και παλιά. Όχι, νομίζω ότι σταθήκαμε εξελικτικά απέναντι στο νέο κείμενο. Υπήρξαν ορισμένα σημεία όπου συζήτησα με τον αρμόδιο της εποπτικής αρχής και μου εξήγησε ότι σε ορισμένου τομεί θέλει περισσότερε αρμοδιότητε και σε άλλου τομεί λιγότερε αρμοδιότητε όταν συνδιαλέγεται με ένα πιστοτικό ίδρυμα. Σε ορισμένες περιπτώσει οι συγκητέ είπαν ότι οι πληροφορίε θα πρέπει να γίνουν δημόσιε άμεσα. Και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να πιστεύουν ότι θα πρέπει να έχουν ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση εφόσον μπορούν να πούν ότι έχω το δικαίωμα να σε υποχρεώσω εσένα πιστοτικό ίδρυμα να δημοσιεύσεις ορισμένα στοιχεία. Και αν δεν μου τα δώσεις τώρα θα σε υποχρεώσω με άλλο τρόπο. Αυτό θέτει τις εποπτικές αρχές σε πολύ καλύτερη θέση θέλουν λοιπόν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτή την ε, ικανότητα, αυτή την εξουσία όχι την υποχρέωση υποχρεωτικά γιατί αυτό μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα αποδοτικό. Κάποιες από τις τροπολογίες μας λοιπόν δίνουν την δυνατότητα όχι να υπάρχει αυτόματη δημοσίευση των δεδομένων από πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά η εποπτική αρχή έχει πλέον την δυνατότητα να συλλέξει τις πληροφορίες αυτές και να τις δημοσιοποιήσει εφόσον αυτή κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Τέτοιου είδους θέματα συζητάμε με το Συμβούλιο και είναι τα θέματα που μου μεταφέρουν οι αρμόδιοι των εποπτικών αυτών αρχών. Ρεκμακ. Ευχαριστώ. Και καταρχάς δεν ζηλεύω τους ηγητές που έχουν όλες αυτές τις ε, τροπολογίες να εξετάσουν. όπως ο κύριος Γκονσιές. Θα ήθελα να σημειώσω τα εξή ότι η εμπειρία που έχουμε από την κρίση είναι ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Καλύτερη επιτήρηση πέραν των συνόρων. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη πάντοτε. Γιατί τον αρχίζουμε να απαγορεύουμε προϊόντα κτλ. θα ήταν Λάθο προσέγγιση θα ήταν ε, να ξεκινάμε, να ξεκινάμε από το τέλο αντί από την αρχή. Α έχουμε πρώτα την κατάλληλη επιτήρηση. Αν εξασφαλίσουμε αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε κερδίσει πολλά και θα, θα είχαμε αποφύγει και πολλά προβλήματα από αυτά που βλέπουμε σήμερα, αν υπήρχε κατάλληλη επιτήρηση. Δεύτερον, πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, απρόσκοπτη λειτουργία των ε, συστημάτων. Έτσι και με μια ρεαλιστική πρακτική προσέγγιση και με την αναζήτηση του τι είναι πραγματικά δυνατό, θα μπορούσαμε να συστήσουμε για μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές αρχές. Αλλά νομίζω πάνω απ' όλο ότι σημαντικό είναι να μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε για μια εθνική αρχή, για τις δράσεις μιας ε, κυβέρνησης κτλ. Και νομίζω ότι όταν έχουμε προτάσεις για πολύ ακραία προϋπόθεση επιτήρησης. Ε, ίσως θα είναι περιβολικό, ξέρετε, πιο, πιο σκόπιμο και φρόνιμο να πούμε ότι εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση, ελέγχεται δηλαδή ότι υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο για κάθε είδου δέσμευση που αναλαμβάνεται έτσι ώστε να, επιλύονται τα προβλήματα. Δηλαδή, τέτοιου είδου κανονισμοί θα μπορούσαν, τέτοιου είδου διατάξει θα είχαν μπορέσει να αποτρέψουν τα προβλήματα στην Ισλανδία, Φερρυπίνο, που υπήρχε πρόβλημα ω προ την επιτήρηση. Αυτό στο λάβουν υπόψη, παρακαλώ, οι συγητές. Κύριος Πόρτας. Ε, são algumas observações muito breves, são até, em alguns Ευχαριστώ πολύ και πολύ σύντομα με κάποιες εμφολίες που έχω να διατυπώσω σε ορισμένες περιπτώσεις. Ξεκινώ με την έκθεση του συναδέλφου Μαργκάιου. Ναι, Θεωρώ σκόπιμη μια κατανομή σε διαφορετικά επίπεδα. Ναι, θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει για κάθε επίπεδο ένα σύστημα εποπτείας. Αλλά όταν αρχίζουμε να μιλούμε για ένα ευρωπαϊκό ταμείο, αρχίζω να έχω τις αμφιβολίες μου. Γιατί αυτό θα απευθυνόταν μόνο σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρουσιάζουν συστημικούς κινδύνους στην Ευρώπη. Άρα θα αποκλείονταν τα μέσου επίπεδου χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό είναι που δεν είμαι σε θέση να καταλάβω. Στην ε, Πορτογαλία, την πατρίδα μου παραδείγματι. Σε περίπτωση απάτης αν πρόκειται για μια τράπεζα που έχει μόνο ένα 2% επί του ΑΕΠ, Μάλιστα, είναι συγκεκριμένη περίπτωση, μια τέτοια μικρή τράπεζα και άρχισε ο Υπουργό των Οικονομικών να λέει ότι δεν, έχει, δεν παρουσιάζει συστημικό κίνδυνο η τράπεζα αυτή. Εν τέλει όμω ε, εθνικοποιήθηκε αυτή η τράπεζα. Και παρόλα αυτά δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν η αλήθεια. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν να γνωρίζουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο ποιες τράπεζες θα καλύπτει. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τα ποσά που θα δεσμεύονται. Εάν αυτά αφορούν μόνο τις πολύ μεγάλες τράπεζες, μπορούν να χρηματοδοτούνται από, την, από τις Τράπεζα. της Με ποιο τρόπο όμως πρέπει να δούμε κάποια μελέτη συγκεκριμένη την οποία θα ζητήσουμε, αλλά θα ήθελα να έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Και τέλει, για να συντομεύω, θα ήθελα για μια φορά να υπογραμμίσω ένα σημείο μιας παρατήρησης κυρίας Γκουλάχ για τη δική της έκθεση ότι βεβαίως και εγώ θα συμφωνούσα στο να είναι η μέγιστη δυνατή η σύγκληση μεταξύ των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών τραπεζών και της εποπτείας. Θα ήθελα να υπάρξει δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία. Αυτό, ωστόσο, ε, σημαίνει μια συνάφεια μεταξύ της μακροοικονομικής εποπτείας και των δομών, πράγμα το οποίο όμως έχει σαν αποτέλεσμα δυστυχώς ότι ε, εισάγουμε πολύ βαριές δομές, δομές δυσκίνητες και ε, αναποτελεσματικές. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος. Σας πω ποιοι είναι οι ομιλητές, Λούλινγκ, Τζούρι. Prezedo wants to come back in again on other things. Pitella. Και μετά θα συνεχίσουμε, θα ξανακούσουμε τους συγγητές. Είμαστε εντάξει. Θα αρχίσουμε, ανοίξουμε και νέο κατάλογο. Παρακαλώ, κυρία Βόρτμαντ Κόλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω με δύο παρατηρήσεις όσον αφορά την έκθεση του συναδέλφου Γκαρσία Μαργάλο για την εποπτεία τραπεζών. Και όπως και την προηγούμενη φορά θέλω και εδώ να μας ενθαρρύνω για περισσότερη φιλοδοξία να εμείνουμε σε αυτά που ζητάμε. Και ο κύριος Σκίνερ και άλλοι είπαν ότι μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε το Συμβούλιο να κουνηθεί. Και είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να τα κρατήσουμε όλα όσα θέλουμε, να κάνουμε το Συμβούλιο να προχωρήσει. Θέλω λοιπόν να πω όπως και ο προλαλής σας, ότι όταν πρόκειται για την εποπτεία των τραπεζών και για κεντρική εποπτεία, σίγουρα πρέπει να υπάρχει <clears throat> και ένα σύστημα ευρωπαϊκό κόστος. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει μόνο η εποπτεία, θα πρέπει να φροντίσουμε και τα κράτη-μέλη. Η αρχή δηλαδή, η νέα, η εποπτική, θα πρέπει να έχει καλή συνεργασία με τις χώρες. Τώρα έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο, το χρηματοδοτούμενο με σφορές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εγώ πιστεύω ότι στα πλαίσια αυτών των καθητήριων γραμμών το Συμβούλιο πρέπει να δεχθεί τις προτάσεις μας. Μια δεύτερη γενική παρατήρηση που έχω να κάνω έχει να κάνει με το πακέτο των ε, Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Οι εποπτικές αυτές αρχές πρέπει να ελέγχονται, προσπαθούν να πετύχουν τη σταθερότητα τιμών. Έχω την αίσθηση ότι διευρύνουμε πολύ τις αρμοδιότητες τελικά των Ευρωπαϊκών Αυτών Επαπτικών Αρχών δεν πρέπει να παραλείψουμε με τίποτα να μιλήσουμε για τη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ίσως μερικά πράγματα πρέπει να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για την έκθεση της κυρίας Γκίκολτ, που είμαι σκιώδης εισηγήτρια από ΤΑΛΚ, συμφωνώ για αυτά που λέει για περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης. Για τον περιορισμό των ρητρών και να μην ακολουθήσουμε τις βρετανικές επιθυμίες σε αυτό το σημείο. Συμφωνώ μαζί της. Αλλά υπάρχουν δύο πράγματα που θέλω να διασαφηνίσω. Από την πρότασή σας που μιλάτε για την απαγόρευση ορισμένων προϊόντων. Και διμερώς το έχουμε συζητήσει. Και εγώ επιμένω να βρεθεί μια λύση. Γιατί δεν έχει να κάνει αυτό τόσο με ένα προϊόν αυτό καθε αυτό, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν αυτό. Αυτό είναι που προκαλεί αστάθεια στην αγορά και όχι το προϊόν αυτό καθε αυτό. Δεν είναι ζημιογόνο, δεν είναι βλαβερό από μόνο του. Και αυτό θα πρέπει να το λύσουμε με διαφορετικό τρόπο και όχι με την ε, απαγόρευσή του. Θα ήταν αυτός καλύτερος δρόμος για να ακολουθήσουμε. τέλος να μπορούν να προσφεύγουν ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές κατά ενός εθνικού συστήματος. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Αυτά είχα να παρατηρήσω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Mrs. Lulling. Η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τους συστημικούς κινδύνους. Και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ουσίας και όχι τόσο να διατρέξω τις διάφορες τροπολογίες που έχουμε εδώ. Η κυρία Γκουλάρ δεν είναι ανάμεσά μας, έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, εγκρίνω κάποιες από τις προσπάθειες αυτές, εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα, με καινοτόμο τρόπο. Αλλά το Συμβούλιο δεν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες πλέον και γι' αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο να, εκφέρει, να φέρει προς τα έξω τις φιλοδοξίες του και συμφωνώ σε αυτά τα οποία λέει η κυρία Γκουλάρ. Η κυρία Γκουλάρ θέλει να υπάρξει διεύρυνση της εκπροσώπησης ε, στα πλαίσια της Επιτροπής Αξιολόγησης Συστημικών Κινδύνων δεν είμαι εναντίον σε επίπεδο αρχής αυτής της διεύρυνσης της παρουσίας και εφόσον όλοι πιστεύουν το ίδιο πράγμα, σίγουρα ε, ε, αυτό δεν είναι πάντα θετικό. Η τάση προς, προς τη διαφάνεια θα έλεγα και προς το άνοιγμα είναι της μόδας, αλλά θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ σοβαροί και οι φιλοδοξίες αυτές θα πρέπει να είναι θα έλεγα κάπως μετριοπαθείς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σίγουρα στα πλαίσια αυτού του νέου οργάνου δεν θα πρέπει να είναι ηγεμονική, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο, να έχει αυτό που λέμε στις εταιρείε μια ελεγκτική πλειοψηφία. Έχει μια αντίληψη γύρω από τα πράγματα αυτά συνολική και έχει αποδείξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη σοβαρότητά της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από ό,τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η φιλοδοξία αυτή περνάει νομίζω με τη χρήση περισσότερο της κοινοτικής μεθόδου και λιγότερο της εθνικής ή της διακυβερνητικής. Πάντως η Επιτροπή αυτή η αξιολόγηση συστημικού κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τραπεί σε μηχανισμό, να μετατραπεί σε μηχανισμό αντίπαλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό θα είναι πάρα πολύ κακό να υπάρξει δηλαδή ανταγωνισμός ανάμεσα στα όργανα, θα ήταν επικίνδυνο και βλαβερό. γιατί η ευρωπαϊκή μορφή εποπτείας είναι έτσι κι αλλιώς διασπασμένη και αυτό δεν είναι καλό. Έρχομαι τώρα στην έκθεση Ντελαροζιέρ που είναι η βάση πάνω στην οποία εργαζόμαστε. Συμφωνούμε όλοι γύρω από τη βάση αυτή. Το θέμα είναι λοιπόν να προσπαθήσουμε με ευέλικτο τρόπο να λιάνουμε τις διαφορές μας. Αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι μαξιμαλιστικές τότε όλα θα πρέπει να τεθούν εκ νέου σε συζήτηση. Η μικροεποπτεία θα πρέπει να είναι εθνική, η μακροεποπτεία θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και αν πραγματικά αυτή την ισορροπία την κλονίσουμε τότε αμφισβητούμε το σύνολο της πρότασης. Συμπερασματικά, εγώ δέχομαι ένα μετρημένο άνοιγμα αυτή της αρχής εποπτείας, αλλά όχι αυτό το οποίο προτείνουν οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι. Υπάρχει μια κίτρινη γραμμή, την οποία δεν θα πρέπει να διανύσουμε. Και εκεί βασίζονται σε αυτή τη λογική και οι τροπολογίες τις οποίες κατέθεσα. Δεν έχουμε αιμονές, κανένας δεν θα μας κατηγορήσει γι' αυτό, αλλά ελπίζω ότι η κυρία Γκουλά θα λάβει υπόψη την άποψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Επιτρέψτε μου να πω ένα πράγμα ακόμα για την έκθεση Μαργκάγιο, Πρόεδρε. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι για μένα κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ να υποστηρίξω τις εκθέσεις Γκίγκολντ και Σκίνερ. Η έκθεση όμως του εξαιρετικού συναδέλφου του Γκαρσία Μαργκάγιο που ζητάει να υπάρξει η λήψη αποφάσεων με την πλειοψηφία, με ενισχυμένη πλειοψηφία, ευνοεί τα μεγάλα κράτη-μέλη εις βάρος των κρατών μελών, των ενδιαμέσων που αποτελούν τα δύο τρίτα των 27. Και σε όλες τις αποφάσεις ε, που έχουν σχέση με τον τρόπο επικοινωνίας αυτών των δύο κατηγοριών, εγώ θα προτιμούσα με τη λογική μία χώρα, μία ψήφος. Βέβαια θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο διαφορετικές κατηγορίες και γι' αυτό θα υποστηρίξω την ισορροπία που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Γκίγκολντ και ο Σκίνα. Και δεν θα συμφωνήσω κύριε Μαργκάγιο με τη δική σας τροπολογία υπαρίθμη 130. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμερίζομαι τις απόψεις κυρία Ζούλη, σε μεγάλο βαθμό. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν την αρμοδιότητα για την νομοθετική ρύθμιση των, ε, της επιτήρησης της εποπτείας. Ήταν πολύ δύσκολη όμως η λήψη αποφάσεων ε, συνέτικων σε επίπεδο Συμβουλίου και τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν τυχόν κατατεθούν, θα κινδυνεύουν να διαταράξουν την ισορροπία στο Συμβούλιο, τις λεπτές αυτές ισορροπίες. Δηλαδή, ίσως να καταστήσουν πιο δύσκολη την εξέβρεση λύσης μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών μελών. Εγώ έχω ζητήσει την απόψη του Υπουργείου των Οικονομικών της Εθνικής Τράπεζας, της, κρατικής, μάλλον, της Κεντρικής μάλλον, Τράπεζας της Σλοβακίας, που λίγο πολύ μου λένε το ίδιο. Όπως άλλωστε πιστεύω θα λένε όλες οι μικρότερες χώρες. Ότι δηλαδή κοιτούν κάποιες βασικές πτυχές της νομοθεσίας τους και την ε, αναθεωρούν. Καλό είναι βέβαια να συζητούνται όλε τι προτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά α είμαστε και ρεαλιστέ. Θα τι απορρίψουν τα κράτη-μέλη. Δεν θα υπησέλθω σε προστασίες λεπτομέρειε, αλλά τα κράτη-μέλη θα θεωρήσουν την ε, στάση μας αυτή ως μια αδικαιολόγητη παρέμβαση εσωτερικά τους. Και όχι μόνο δικαιολόγητη, αλλά και απρόσφορη. Η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, κατά την άποψή μου, δεν είναι ζήτημα φιλοδοξίας. Πρέπει να διαχωρίσουμε τις φιλοδοξίες μας από την πραγματικότητα. Και την πραγματικότητα να τη συζεύξουμε με τις ευθύνες που φέρουμε. Βλέπω λοιπόν στο μέλλον επιφυλάξει από πλευρά των ε, οργάνων της, ε, του κράτους Σλοβακίας και φαντάζομαι ότι όλα τα κράτη-μέλη θα θέλουν να διατηρήσουν τις εποπτικές τους εξουσίες οι εθνικές αρχές. Δεν θα συμφωνήσουν δηλαδή να έχουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της ε, μετατόπισης εξουσίας μας στην Ευρώπη ως προς εθνικές τους αγορές και ως προς τα δημοσιονομικά ζητήματα το Δεκέμβριο το ΕΚΟΦΗΝ συμφώνησε σε ένα πλαίσιο για την επίλυση των διαφορών μεταξύ ποπτικών αρχών και για να προχωρήσω σε κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με μια απλή πλειοψηφία του ενός μέλους, της μιας ψήφου μάλλον ένα μέλος, όχι με ειδικέ πλειοψηφίες στο Συμβούλιο. Αυτή είναι η ιδέα στην οποία ίσως να συγκρουστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχε περιπτώσεις. θα προσπαθήσω να συνοψίσω μέσα σε ένα κείμενο και ένα λόγο θα τις θα αποστείλω στον καθησυγητή. υπάρχει επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από ό,τι βλέπω τα μικρότερα μάλλον, αλλά και κάποια μεγαλύτερα κράτη, δείχνουν μια μάλλον σταθερή στάση απέναντι στην υπόθεση Αυτό όσο το βλέπουμε και σε επίπεδο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ε, ζητήσω να λάβετε υπόψη σας τις τροπολογίες που καταθέσαμε με διάφορους συναδέρφους και που έχουν να κάνουν με τρία θέματα κυρίως. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία των αρχών αυτών. Δεύτερον, να ενισχύσουμε την αντιπροσωπευτικότητα ε, των αρχών αυτών. Και τέλος, θέλουμε το Κοινοβούλιο να έχει μια ισχυρή θέση απέναντι στις αρχές αυτές. Τώρα θα μπω στις λεπτομέρειες και θα περιγράψω ποιες είναι οι τροπολογίες μας. Για μία από τις αρχές αυτές, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ενίσχυση της εκπροσώπησης ορισμένων χωρών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με άλλα λόγια, θα θέλαμε εκπροσώπους και από τις νέες και από τις παλιές χώρες μέλη. Όταν τώρα μιλάμε για ανεξαρτησία, ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη η οποία φροντίζει για το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν χρειάζεται η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι θα είναι πιο ανεξάρτητες οι αρχές αυτές, κατά τη γνώμη μας. Έρχομαι τώρα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ θα θέλαμε να έχει λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλω τώρα να μιλήσω λίγο για το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Το συζητήσαμε λιγάκι και χθες που είχαμε εδώ τον κύριο Τρισέ. Η αρχική πρόταση δεν μιλάει ρητά για την σύνθεση της Steering Committee. Η πρότασή μας είναι να πούμε δυνατά και ξεκάθαρα ότι εκπρόσωποι και μέσα και εκτός Ευρωζώνης πρέπει να συμμετέχουν στην Επιτροπή αυτή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα θέλαμε να συμμετέχουν στις δράσεις των αρχών αυτών. Η υποχρέωση των αρχών αυτών να λογοδοτούν πρέπει να διατυπώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην οδηγήσει υπερβολική γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αφήνω τους συζητητές για το τέλος. Ο κύριος Πιτέλα έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η διαρκή δεν έχει ξεκινήσει μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Καλό λοιπόν θα ήταν να έχουμε μία θέση σαφή εμείς μέσα στο Κοινοβούλιο, μια θέση που να υιοθετούν οι πάντες και νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό εκφράζουν οι παρεμβάσεις. Κοινή λοιπόν στάση αλλά χωρίς υποχωρήσεις ότι έχουμε να κάνουμε μεγάλα, μεγάλες προκλήσεις και σοβαρά διακυβεύματα. Εάν υποχωρήσουμε, το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να προδώσουμε τον πολίτη. Όποιος δεν θα καταλάβει γιατί ε, υιοθετεί τόσο ασθενική στάση απέναντι στο Συμβούλιο, το κοινοβουλίο μας. Τώρα να σας πω πολύ γρήγορα ποια είναι τα κεφάλαια στα οποία ε, αναφέρονται οι 90 μου τροπολογίες. Πρώτο σημείο, τα θέματα της εκχώρησης ε, αρμοδιοτήτων και της επιτροπολογίας με τροπολογίες που στόχο έχουν ε, να μην μπορεί να τροποποιήσει τις τεχνικές ε, διατάξεις ή προδιαγραφές που θα έχει υιοθετήσει η Εποπτεύουσα Αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τον προσδορισμό του πώς θυμάται ο συστημικός κίνδυνος και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών. Για τους ίδιους λόγους είμαι και θετικά δικαιμένος απέναντι σε μία απόφαση της Επιτροπής δεσμευτική για τις αρχές στις οποίες απευθύνεται απόφαση η οποία θα εξασφαλίσει και την ασφάλεια του δικαίου στους κανόνες της επιτήρησης υποπτίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι θα, καλύπτει, θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε ε, ασυνέπεια ως προς την τήρωση των ευρωπαϊκών διατάξεων. Στη συνέχεια ζητούμε μεγαλύτερη προστασία, σαφέστερη προστασία των επενδυτών θα έπρεπε να είναι ο κύριος μας στόχος και ένα πιο σαφώς προσδιορισμένο ρόλο της ομάδας των εμπλεκομένων φορέων, των ενδιαφερομένων φορέων. Για δε την ε, δυσφαιριστική ρήτρα, το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αφηρημένη υπερβολικά ε, γενικόλογη περιγραφή της ευθύνης των κρατών που θα μπορούσαν ακόμη και να οδηγήσουν σε παράλυση της δραστηριότητας της ε, αρχής. Για να κλείνω λοιπόν διαφάνεια, έλεγχο στον τομέα των παραγόγων, στα χέρια της Επιτροπής Εποπτείας. Ευχαριστώ Ελίσσα Φεραίρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Και είναι σημαντικό να υπάρξει πλήρης συνοχή στις διάφορες, μεταξύ των διαφόρων αρχών. Και μια που συμμετέχω στο Cross Border ε, Banking Resolution, προσπαθώ να καταλάβω τις λεπτομέρειες της τελικής πρότασης που θα υιοθετήσει ο κύριος Μαργάγιο. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα ειδικό σύστημα για τις τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όμως σιγά σιγά θα διευρυνθεί και θα συμπεριληφθούν και τα διασυνοριακά ιδρύματα. Έτσι δεν είναι. Ή θα διατηρήσουμε τα τρία συστήματα χωριστά Ισαΐ. Δεύτερον. Για το Ταμείο. Συμφωνώ με τις φιλοδοξίες που έχουμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο χρηματοδοτούμενο με συγχωρές χρηματοπιστωτικών ιδρωμάτων. Εγώ πιστεύω ότι το Ταμείο έχει νόημα εφόσον είναι ο κλάδος που προστατεύει από τον κίνδυνο. Στην ίδια την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα υπάρχει μια task force και ο στόχος του Ταμείου συμπεριλαμβάνει και την προστασία των ε, πιστωτών ή μόνο του συστήματος από συστημικό κίνδυνο. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι να πούμε σαν είδα σωτηρίας για τις τράπεζες και άλλο είναι περιορίζουμε τη ζημιά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ξέρω περισσότερα για το ταμείο αυτό. Τρίτο, όταν παρεμβαίνει το ταμείο σε μια συστημική τράπεζα, πρέπει να παρεμβαίνουμε με ένα σύστημα, όχι με διαφορετικά νομικά συστήματα. Οπότε, πώς θα γίνει αυτό. Θα φτάσουμε σε κάποια μεγαλύτερη εναρμόνιση. Υπάρχει μια αμφιβολία για το νομικό σκέλος εδώ που δεν είναι εντελώ ξεκάθαρο για μένα. Αλλά θα μου το εξηγήσετε, είμαι σίγουρη. Όσον αφορά τις εισφορές στο Ταμείο, δέχεστε ότι πρόκειται για εισφορές που βασίζονται στον κίνδυνο, ανάλογα δηλαδή με τον κίνδυνο. Θα δούμε τι λέει η Βασιλεία ή όχι. Και κάτι ακόμα γι' αυτό. Στην περίπτωση της Ισπανίας σήμερα δημιουργούνται εθνικά ταμεία όπως στην Ισπανία. Οι χώρες όμως έχουν και συστημικές επιχειρήσεις. Εσείς πώς βλέπετε την μεταβίβαση από την εισφορά ε, στα εθνικά ταμεία σε εισφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Πώς θα γίνεται η διάσωση με ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο. Πάντως η διάβρεση πρέπει να γίνει. Αν θέλουμε μια ευρωπαϊκή αγορά πρέπει συγχρόνως να έχουμε κάτι τέτοιο όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Δεν πρέπει να χαθούμε στις λεπτομέρειες. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας μετά. Ευχαριστώ. Case Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμείς προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μια συνεπή γραμμή, όπως όλες οι ομάδες, μεταξύ των τριών ε, προοπτικών αρχών και του Ταμείου Συστημικών, ε, ε, της Επιτροπής Συστημικών κινδύνων. Αυτό που θέλουμε είναι με τους εισηγητές μας να διατηρηθεί η κοινή γραμμή για όλες τις εκθέσεις, να μην αρχίσουν οι αποκλήσεις που διαφαίνονται τώρα. Υποστηρίζουμε την θέσπιση των νέων αρχών και της Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου, την ε, σύσταση, την εκπόνηση και την ε, υιοθέτηση ενός κοινού ε, συνόλου κανόνων, ενό κοινού κώδικα κανόνων. Θα πρέπει όμως και εγκαίρως να συσταθούν όλα αυτά και οι εκθέσεις να παραμένουν όσο δυνατόν πιο απλές στο τωρινό στάδιο. Είναι πολλά τα εμπόδια που έχουμε να ξεπεράσουμε και όπως σας ανέφερα και νωρίτερα σε άλλες ακροάσεις, μπορεί το Ταμείο να έχει κάποιο λόγο ύπαρξης, αλλά χωρίς ε, κατάλληλη μελέτη, τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα διατεθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Και επίσης οι ρυθμιστικές αρχές συμφωνούν όλες ότι την καλύτερη ρυθμιστική λειτουργία μπορούν να την έχουν σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο οι ρυθμιστικές αρχές. Υπάρχει το ε, κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να λάβουν αυτή τη δραστηριότητα αμέσω και γι' αυτό προτιμούμε όπως ο Πίτερ Σκίνερ την εξέλιξη και όχι την επανάσταση. Ας αρχίσουν να λειτουργούν αυτές οι αρχές, να αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά τους προβλήματα και μετά να δούμε αν θα τους δώσουμε και περισσότερες εξουσίες. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, την προηγούμενη εβδομάδα μου είπε κάποιος ε, στη συνεδρίαση εδώ ότι, το όνομα, ότι ο τίτλος ομάδας μου ECR τώρα πια δεν σημαίνει συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές αλλά Συμβούλιο των ε, εκπρόσωποι του Συμβουλίου ECR, Council Representatives. Όχι, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Απλώς θεωρώ ότι είναι καλύτερο να δώσουμε τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό και την υποδομή σε αυτές τις εποπτικές αρχές για να λειτουργήσουν σωστά το ταχύτερο δυνατό. Και μετά να κοιτάξουμε εάν θα διευρύνουμε τις αρμοδιότητές τους. Παρακαλώ λοιπόν. Θέλετε να σημαίνει κάτι άλλο για λίγο το ε, ακρονίμιο της ομάδας μου. Έστω, αλλά κάντε μια προσπάθεια για να περάσουμε στην πρώτη ανάγνωση της πρότασης. Γιούργεν. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σκιώδης ηγητής. Ο Τόμας Χέντλ έχει αυτή την αρμοδιότητα μου, αλλά δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Και έτσι με παρακάλεσε να μιλήσω εγώ εκ μέρου του. Αν μου επιτρέπετε. Οι δικέ μα τροπολογίε ιδιαίτερα ζητούν την ε, μπλοκή των, ε, της κοινωνίας των πολιτών στις εποπτικές αρχές τα συνδικαλιστικά σωματεία που έχουν ε, και την ανεξαρτησία και την ε, πραγματογνωμοσύνη και πιστεύουμε ότι χωρίς τη δική του συμμετοχή δεν θα, μπορούσαμε, δεν, θα μπορούμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε και να ελέγξουμε τις κρίσεις όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. Χρειάζεται λοιπόν η παρουσία τους και ο έλεγχος τους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της παρακολούθησης της ε, δράσης αυτών των αρχών και σε συνδυασμό με τις ε, δράσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι δομές είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, εν μέρει έχω καλυφθεί πρέπει να δούμε εάν έχει νόημα να τις αναπτύξουμε τις αρχές αυτές σε τρεις διαφορετικούς γεωγραφικούς, σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Και επίση θέλω να πω ότι συμφωνούμε με τον Σβέν ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτέ οι αρχέ να απαγορεύουν τα επικίνδυνα ή τοξικά, όπω λέγονται, χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και ο συνάδελφο Λαμπέρ το είχε πει πριν από κάποιε συνεδριάσει, δεν μπορώ πρώτα να τον υποστηρίξω. εν ολίγης είμαστε υπέρ της απαγόρευσης όποιων επικίνδυνων ε, προϊόντων εντοπίζει το Συμβούλιο. Χρειάζεται νομίζω αυτή η διάσταση για την ε, σωστή ε, ρύθμιση. Αυτά μου είχε ζητήσει να πω ο Τόμας. σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Right. Uh, I'm now moving back to the rapporteurs. So those... Επιστρέψουμε. Επιστρέφω στους εισηγητές. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν να σχολιάσουν αυτά που άκουσαν. Πρεσέδω. Ευχαριστώ. Με βάλατε στην αρχή. Ναι. Αλλά εγώ δεν έχω να κάνω σχόλια για τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Δεν νομίζω ότι άμεσα σε μένα απευθύνθηκε κάποια ερώτηση. Θέλω όμως να αποφεληθώ λίγο ε, από την ευκαιρία για να μιλήσω ως συντάκτης τροπολογίας ζήτησα τροπολογίες και στις τρεις εκθέσεις, γιατί θέλω να πάνε πιο μακριά από την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επέβαλα λοιπόν τροπολογίες στις τρεις ε, ε, εκθέσεις προς την ίδια κατεύθυνση και ίσως ευρύτερα στην έκθεση Γκαρθία Μαργάγιο, που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και γιατί, να σας πω, μ' αρέσει η μουσική, αλλά θα μπορούσαμε να πάμε περισσότερο σε βάθος. ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία διαλόγου που θα έχουμε με το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκινήσει από μια πολύ στέρεα βάση και με σαφείς στόχους. Η βιωσιμότητα είναι ένας από τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε με την εποπτεία. Δεν είναι αυτός σκοπός όμως. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που είναι η σταθερότητα, μακροπρόθεσμα, η σχέση των δημοσιονομικών με την πραγματική οικονομία. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν έναν κοινό παρονομαστή σε όλες τις προτάσεις. Πρέπει επίσης να δούμε τι ακριβώς είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δημοσιονομικής Εποπτείας και αυτό να το κάνουμε όχι απλοϊκά. Υπάρχει για τις μεγάλες τράπεζες, μα μέσα σε αυτές τις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν και άλλες μικρές, που πρέπει και αυτές να εποπτεύονται σε εθνικό επίπεδο. Πώς διαρθρώνεται αυτή η ευρωπαϊκή εποπτεία λοιπόν με τα εθνικά συστήματα εποπτείας. Εγώ θεωρώ ότι κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν πρέπει να είναι κάτω από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Να βάλουμε δηλαδή ένα κατόφλι κάτω από το οποίο δεν πρέπει να είναι κανείς. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκό δημοσιονομικό χώρο. Έπειτα να έχουμε ένα οριζόντιο και προδευτικό σύστημα. Αυτά ζητάω με τις τροπολογίες μου. Υπάρχει μια πτυχή πολύ σημαντική νομίζω και είναι να αποφύγουμε να έχουμε καθαρά τεχνικού χαρακτήρα ρύθμιση. Η Βασιλεία όταν μιλούσε για τραπεζική εποπτεία έλεγε ότι πρόκειται για εφαρμογή του νόμου, αλλά πρόκειται επίσης και για ασφάλεια και για φερεγγιότητα. Εμείς λοιπόν αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δούμε πρώτα απ' όλα ποιε είναι οι πτυχέ τη φερεγγιότητα και τη σταθερότητα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εποπτεύονται από ευρωπαϊκό επίπεδο. Έπειτα ο συστημικός ε, κίνδυνος και ο διασυνοριακός κίνδυνος. Εδώ υπάρχουν ορισμοί που μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής εποπτείας. Θέλουμε να υπάρχει συνοχή, να είναι αποτελεσματική υποπτή αυτή. Τι σημαίνει single rule book. Έχει οδηγίες που κανείς δεν καθόρισε και εμείς πρέπει να πούμε τι σημαίνουν. Εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει εμείς να πούμε τι ακριβώς είναι αντικείμενο νομοθεσίας, και τι είναι αντικείμενο πράξης ε, εξουσιοδότησης. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε. Να βασιζόμαστε όχι μόνο στην ομοθεσία αλλά και στην αξιολόγηση κινδύνου και να φτιάξουμε ένα κατάλογο. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι το εξής. Η τραπεζική αρχή εφόσον κάνει άμεσα εποπτεία Είναι πολύ σημαντικό τις αρμοδιότητες αυτές να τις ορίσουμε και να φροντίζουμε να υπάρχει ασφάλεια. Ελπίζω αυτά να λυθούν στο μέλλον. Πιστεύω επίσης ότι οι αρχές πρέπει να είναι περισσότερο ισχυρές και ανεξάρτητες. Και όταν πρόκειται για τεχνικούς κανόνες, για τις κατεξουσιοδότηση πράξη, να υπάρχει εποπτεία όπως και οι εθνικές αρχές πρέπει να κάνουν τέτοια εποπτεία και ο ρόλος να είναι δεσμευτικός. Οι αποφάσεις, ε, οι συστάσεις να είναι δεσμευτικές. Οι δημοσιονομικές αρχές εξαρτάται από το μέγεθός τους και εξαρτάται αν μιλάμε για επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο εμπιστεύομαι τον εισηγητή για τα εξή. Πρώτον, η άμεση εποπτεία και το Ταμείο Οικονομικής Προστασίας. Εντάξει, δεν με ενοχλεί η ιδέα μιας άμεσης εποπτείας. Άμεσης, άμεσης. Απευθείας. Από της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πρέπει να υπάρχει εδώ συνοχή. Πού θα γίνεται η άμεση εποπτεία. Έχουμε τις 25 τράπεζες που είναι πάνω από 40% του ενεργητικού στον κόσμο. Ποιος θα δικάνει κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Εγώ θα ήθελα αυτό να γίνεται διμερός. Και όχι γιατί θέλω να αναβάλω το θέμα, Ισαΐ, αλλά γιατί υπάρχει μια συμφωνία στο Λονδίνο, μιλήσαμε για εντοπισμό των ε, ιδρυμάτων των πιο μεγάλων. Πιστεύω λοιπόν καλύτερα να γίνει διμερός και όχι πολυμερός η άμεση αυτή εποπτεία. Και αν δεν το θέσει κανένας άλλος, να το θέσουμε εμείς. Τέλος, να πούμε ποιες είναι οι τράπεζες στις οποίες πρέπει να γίνεται εποπτεία. Τέλος, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Οικονομικής Προστασίας, συμφωνώ με αυτά που είπε η Λίσσα Φερέιρα. Ο κίνδυνος είναι να γίνει από ορισμένε τράπεζες, να μην έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα διαρθρώνεται με ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου. είναι ένα ζήτημα που αν μη τι άλλο πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Γκαρθία Μαργάγιο είναι εισηγητής με μεγάλη εμπορία, εμπειρία, οπότε βασίζομαι σε αυτόν. Εδώ πρέπει να ψηφίσουμε, οπότε να έχουμε και τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Ο κύριος Μαργάγιο τότε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω πολύ σύντομα σε όλους σας. Και θα ξεκινήσω με τον κύριο Σκίνερ. Όπως και η συντηρητική θέλει μια εξελικτική διαδικασία και όχι μια επανάσταση. Το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε για να αλλάξουμε ή να αλλάξουμε χωρίς να αλλάζουμε τίποτα. Ε, ως φίλος μου έδωσε την... μου είπε ότι η ιδέα αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά ως Άγγλος, μου είπε, μιλάω ως Άγγλος τώρα, πρέπει να περιμένω. Ως φίλος ναι, ως Άγγλος να περιμένουμε. Για το ταμείο. Τα στοιχεία δεν είναι ακριβώς αυτά που έχω. Σε μια εφημερίδα διάβασα ότι το ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο για τις τράπεζες. Αλλά τα νούμερα που έχω εγώ από τον ίδιο των κλάδων λέει ότι η απόλυση των ασφαλιστικών εταιρείων ήταν το ένα έκτο από εκείνο απόλυση τραπεζών. Και το κεφάλαιο που ζήτησαν ήταν το 1 ένατο από εκείνο που ζήτησαν οι τράπεζες. Αυτές είναι οι διαστάσεις του προβλήματος, έτσι, για να συγκρίνουμε ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Τώρα μπορεί δεν υπάρχει κάποιος που θα πει κάτι άλλο. Ο κλάδος λέει ότι υπήρξε συστημικός κίνδυνος στις εταιρείε εκείνες που είχαν περιορισμένε τραπεζικές δραστηριότητες ε, από την Ολλανδία για παράδειγμα και ασφαλιστικέ εταιρείε το αρχικό πρόβλημα ήταν στο Λονδίνο, δεν ήταν ε, ούτε στην Αμερική ούτε αλλού. Και τέλος, μιλάει για τα monoliner. Και έχω εδώ πέρα τα στοιχεία και τα ονόματα που είναι στη διάθεσή σας, μπορώ να σας τα δώσω κάποια άλλη στιγμή. Για την κυρία Βίκη Φόρτ μου λέει ότι συμφωνούν με το Συμβούλιο. Είναι προφανές. Το Συμβούλιο έχει εξαντλήσει την πρόταση της Επιτροπής που μιλάει για την έκθεση Λαροσιέρ, η οποία η ίδια η έκθεση Λαροσιέρ λέει δεν πήγε πιο μακριά γιατί έπρεπε να δει πρώτα αν αυτές οι προτάσεις θα γίνουν αποδεκτές. Το Συμβούλιο τι θέλει. Θέλει να μειώσει τις ε, εξουσίες της Ευρωπαϊκή Αρχές και βάζει και μια ρήτρα που είναι το opt-out το αγγλικό που λέει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από τους ομοτήμους του στο Συμβούλιο αν πιστεύει ότι μια απόφαση ε, το πλήττει δυσημονιωμικά και εδώ είπε ο κύριος Λαροσιέρ. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή αυτή να το διευκρινίσει παρετέρω. Ο κύριος Χάρτμακ αναφέρεται στις αιτίες της κρίσης και στα μαθήματα της κρίσης. Έχουμε την έκθεση Λάροσερ και την έκθεση Τέρνερ. Ο Τέρνερ βασίζεται σε δύο παραδείγματα. Λέμαν και η Ιρλανδική περίπτωση οι ασφαλιστικές εταιρείες βασίζονται στην περίπτωση της CG. Αλλά εγώ περιορίζομαι στο Λέμαν και στην Ισλανδία. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Μόνο δύο. Ή που δίνουμε περισσότερες εξουσίες στην εποπτεία της αφιτρίωνας χώρας, που μπορεί να απαγορεύσει μέσω θηγατρικών να γίνονται δράσεις, που λέει ο κύριος Στάρνερ σημαίνει ότι σταματάμε με το ευρωπαϊκό διαβατήριο και με την ιδέα μιας εσωτερικής αγοράς ε, δημοσιονομικών ε, προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή έχει δύο σκέλη. Είναι το Συμβούλιο Εποπτών που μπορεί να παρετηθεί σε περίπτωση διαφωνίας αν δεν κάνουμε τίποτα, μπλοκάρεται το θέμα και δεν υπάρχει λύση ή Πάμε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που της δίνουμε την εξουσία διαμεσολάβησης δεσμευτική και που μπορεί έτσι να υποχρώσει να προχωρήσουμε ε, σε κάποιες δράσεις. Ο Όρουελ έλεγε ότι όλοι είμαστε ίσοι, αλλά μερικοί είμαστε πιο ίσοι από τους άλλους. Και η πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχουν ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πρέπει να σώσουμε, όπως το είδαμε στην περίπτωση Λέμαν, γιατί αν πτωχεύσουν, τότε δημιουργούν μια γενικευμένη κρίση με μεγαλύτερη ανεργία, με μείωση της ανάπτυξης κτλ. Ωραία. Ποιος προσέχει όμως, ποιος εποπτεύει τα πράγματα και ποιος πληρώνει τα σπασμένα. Εγώ λέω ότι στην περίπτωση που κάποιος πρέπει να εποπτεύσει είναι η τραπεζική αρχή εξορισμού επειδή είναι υπερεθνική η καλύτερη περίπτωση οι τοπικές αρχές από όταν χάνουν. Το είδαμε. Στην περίπτωση των αποταμιευτών. Στην Αγγλία, Φλανδία κλπ. Αν λοιπόν την ευθύνη για την εποπτεία τη δώσουμε λοιπόν όπως είπαμε το σημαντικό είναι ο κίνδυνος όχι η διάσταση, όχι ο διασυνοριακός χαρακτήρας ούτε τα άλλα κριτήρια τα οποία υπάρχουν και μπορούμε να προσθέσουμε κάποια. Τα θύμισε και ο κύριος Πρεσέδο είναι λίγα. Ο συντονιστής, ο εισηγητής από τους συντηρητικούς είχε πει ότι αν υπήρχε ένα ανώτερο επίπεδο εποπτείας δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το πρόβλημα. Τώρα έχουμε στο δεύτερο. Ποιος πληρώνει? Μα θα προσπαθήσουμε χρησιμοποιώντας τα λόγια του Ομπάμα, δεν θα βάλουμε τη Wall Street να πληρώσει τη Wall Street. Το είπε και ο Σάντσες Πρεσέδο. Και το λέει και η στρατηγική 2020 που λέει ότι πρέπει να ζητήσουμε εισφορές από τα χρεμπιστοτικά ιδρύματα που να είναι κατά πρώτον υπεύθυνα να καλύψουν τη ζημιά. Αυτό τι σημαίνει. Μιλάμε για ε, ομόλογα στην περίπτωση για παράδειγμα της Ελλάδας. Ναι, αλλά είναι πολύ αργά τώρα να φτιάξουμε ένα νομισματικό ταμείο. Αλλά τελικά ποτέ δεν φτάνουμε στην ώρα μας. Πάντα κατόπιν εορτής θα θυμόμαστε. Η κυρία Λούλινγκ αναφέρθηκε στην απόφαση. Μια ψήφο ο καθένας. Το συζητάμε. Εγώ είμαι υπέρ του ο καθένας να έχει μία ψήφο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό, γιατί όταν τελικά κάποιος πρέπει να πληρώσει ανάλογα με τις επιπτώσεις στα κράτη-μέλη, δεν ξέρω κατά πόσο τα θα φτάνουν. Πάντως, ευχαρίστως να το συζητήσω. Αυτό που επίσης συζητάω είναι ότι όταν ζητάμε από τους ομότιμους όταν ένα κράτος μέλος λέει «Α, τι είπε η τραπεζική αρχή» δεν μ' αρέσει και πρέπει να είναι οι ομότιμοι στο Συμβούλιο αυτοί που θα αποφασίσουν, αυτό το κράτος μέλος να μην μπορεί να ψηφίσει. Ό,τι πλειοψηφία θέλετε, αλλά να μην μπορεί να ψηφίσει. Και σίγουρα θα με στηρίξουν πολλοί και θα με μισήσουν πολλοί άλλοι. Ε, την κυρία Γιώργη, συμφωνώ. για τις παλιές και τις νέες χώρες. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει να χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία, να πούμε ότι ορισμένες ε, βρίσκονται υπό εξαίρεση, υπό καθεστώς εξαίρεσης και άλλες όχι, αντί opt-out. Αν η Επιτροπή πρέπει να επικυρώσει τις ε, αποφάσεις, αυτό προβλέπει η συνθήκη. Η διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής για να τροποποιήσει μερικώς τις αποφάσεις είναι πολύ μικρή. Για το ρόλο του Κοινοβουλίου συμφωνούμε. Ο Λάσκες δούλεψε με μένα και έκανε κάτι σαν beauty contest. Καλεστία για το ποιοι αρέσουν, ποιοι δεν αρέσουν. Ο κύριος Πιτέλα τώρα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Υπάρχουν δύο τρόποι μόνο για να κάνει κανείς μια έκθεση εδώ ή να προσπαθήσει να πει αυτά που αρέσει το Συμβούλιο για να πειράσει τις αποφάσεις του και να υπάρξει γρήγορα μια απόφαση και να πάρει μετάλλιο ο εισηγητής ή να προσπαθήσει να ανοίξει νέους ορίζοντες σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Γιατί και το Συμβούλιο εξελίσσεται. Το Συμβούλιο για τη Στρατηγική 2020 είπε ότι πρέπει να ζητήσουμε από τον χρηματοπιστικό ε, τομέα να πληρώσει τα σπασμένα και έχει προχωρήσει και αλλάξει και πολύ περισσότερο σε άλλους τομείς. Η καλύτερη στρατηγική για να το πετυχαίνουμε αυτό είναι να πηγαίνουμε με φιλόδοξες προτάσεις, με φαντασία και να στηρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο την συνδιαλλαγή. Ο άλλος δρόμος είναι πιο απλός. Πάντα γίνεται. Αν θέλουμε να παρετηθούμε από κάτι, παρετούμαστε και τελείωσε. Τα λέμε, πίνουμε καφεδάκι μαζί και ξαναγυρνάμε πίσω χωρίς κανένα πρόβλημα και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Για την κυρία Φερέιρα. Μου μιλήσατε για φιλοδοξία, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και εγώ έχω καλά λόγια για σας. Τώρα ρωτάτε ποιες είναι οι αρχές του συστημικού και ποια είναι τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι διεθνή. Είναι το Συμβούλιο της Τραπεζικής Αρχής που αποφασίζει για τα κριτήρια. Για τις εισφορές ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώνει όσο γίνεται λιγότερο για την κακή διαχείριση ε, κάποιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κύριε Σέμπολ, οι συγκητές θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, όσον αφορά εμένα τουλάχιστον, για τον ρεαλισμό, την εξέλιξη κτλ. Κοιτάξτε, όταν συζητήσαμε τη διαδικασία λαμφαλουσία εδώ, λέγαμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει νομοθετικές διαδικασίες, γιατί επιπλέον, γιατί η διαδικασία μέχρι τότε ήταν πολύ ε, αργή για να προσαρμοστεί σε μια με εξέλιξη που είχαμε. Ποτέ δεν ε, κολλησεργήσαμε εμείς. Και μάλιστα είχαμε και έναν επίτροπο για την εσωτερική αγορά και κάθε φορά που του λέγαμε ότι πρέπει να ρυθμιστούν κάποια προϊόντα, τα παράγωγα για παράδειγμα, ή σκεφτόμενοι του κινδύνου ή ότι έπρεπε να υπάρχουν ρήτρε διασφάλιση, μεγαλύτερη εποπτεία ή ότι πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση. Μα έλεγε ότι δεν γινόταν, ότι ήταν πολύ νωρί και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ευτυχώ ο σημερινό επίτροπο φαίνεται ότι ευθυγραμμίζεται πολύ περισσότερο με εμά. Και αυτό με χαροποιεί όλους ιδιαίτερος, όπως φαντάζεστε. Κύριε Κλώτ, συμφωνώ για το θέμα τις τοποθεσίες. Αν θέλουμε αποτελεσματικότητα, όλες οι αρχές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο σημείο, να έχουν το ίδιο προσωπικό και έναν ενιαίο Ευρωπαίο επόπτη. Μετά από αυτά που γίνανε στην Ελλάδα, τώρα λένε ότι φυσικά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, κερδοσκοπικές ε, προσπάθειες που καταλήγουν και φέρνουν την Ελλάδα στην θέση που τη φέρανε. Κύριε Πρεσέντα, θα τελειώσω με εσά. Ευχαρίστω να το βάλω αυτό που θέλετε, όπου θέλετε. Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή σε σχέση με τις εθνικές. Ε, όταν υπάρχει ένας κίνδυνος, οι εθνικές αρχές λειτουργούν κατά εξουσιοδότηση όπως και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Υπάρχουν ε, πράγματα που είναι περισσότερο ευρωπαϊκά ή περισσότερο εθνικά, τα ξέρουμε αυτά. Για την ασφάλεια συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω και το λέω και ισχύει για όλους, είναι ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε κατακαιρματισμό σε θέματα τυποποίησης και ρύθμισης. Ενώ στα κριτήρια και τις πρακτικές εποπτείες μιλάμε για κατακαιρματισμό. Θέλουμε εναρμόνιση των κανόνων, ώστε όσοι δρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε 18.000 διαφορετικά έντυπα, γιατί θέλουμε να ικανοποιήσουμε 27 διαφορετικά καπρίτσια των 27 διαφορετικών ε, χωρών. Και μιλάω για καπρίτσιο, γιατί υπάρχει η θεωρία αυτή ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το κτίριο που θυμίζει το τυρί καπρίτσι 2 που είναι ο βάλου το ίδιο σχήμα και μιλάω και εγώ λοιπόν για τα καπρίτσια των θεών και για το καπρίτσιο πολλών Ευρωπαίων. Σβέν, ύστερα από τόσο μακροσκελή συζητήσει σήμερα, ακόμη και οι βουλευτέ εξαντλήθηκαν. Ορισμένοι πρόσωποι του Συμβουλίου έχουν ήδη αποχωρήσει. Άλλοι είναι ακόμα εδώ μεν. Δεν εννοούσα εσά. Μα είπε του, δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό θα πρέπει να αναπτύξω τα σχόλιά μου. Η Σιλβή λέει όχι σε μεγάλο, μάλιστα. Για την κυρία Λούλινγκ, η οποία επέμενε πω υπάρχει μεγάλη διαφορά ω προ τη διαδικασία των ψηφοφοριών για τροπολογία 130 για την ε, αρχή για την εποπτεία τραπεζών και ότι θα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της εκθέσεως Κίνερ και της δικής μου αφενός και του Χωσέ Μαρία Μαργκάγιο αφετέρου. Εγώ Ξαναδιάβασα πάλι το κείμενο. Ελάχιστε φορέ βλέπω. Δεν βλέπω μεγάλε αποκλήσει, αλλά θα πρέπει να το ξανασυζητήσω με του συναδέλφου. Πέραν αυτού. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν στο μεγαλύτερο του βαθμού τον κύριο Πιτέλα Δεν το είχα υπόψη μου, αλλά είναι μια καλή ιδέα να το συζητήσουμε. Σχετικά με την άμεση επίβλεψη των υπηρεσιών που χορηγούν τα στοιχεία, είναι κάτι πάνω στο οποίο θα συμφωνήσουμε έτσι και αλλιώ. Νομίζω ότι η βασική συζήτηση την οποία θα πρέπει να κάνουμε αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι εκθέσεις αυτές θα αποφασιστεί να είναι απαιτητικέ ή όχι ή πόσο απαιτητικέ θα πρέπει να είναι. Βασική μας γραμμή θα πρέπει να είναι ή τουλάχιστον είναι αυτή τη στιγμή το να μην θίξουμε κάποια προβλήματα τα οποία είναι τέτοιου μεγέθους που θα καθυστερήσουν τη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι βέβαια το οποίο ίσως να μην αρμόζει απόλυτα με το ρόλο του Κοινοβουλίου σε αυτή τη φάση. Στη συγκεκριμένη φάση ε, το, το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να προσβλέπει από τους Υπουργούς Οικονομικών του Συμβουλίου, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να δουν με ποιους τρόπους θα συμφωνήσουν και απλά να διαπιστώσει το τη δημιουργία του προβλήματος εάν τυχόν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στους εμπλεκομένους. Η λύση η οποία θα πρέπει να βγει από τη διαδικασία θα πρέπει να εμπνέεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά της κρίσης των τελευταίων χρόνων και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την γνώση που έχουμε σωρεύσει από τις αποτυχίες και τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων. Αν σαν παράδειγμα έχουμε κάποιες ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ασκείται και από ποιους θα ασκείται η εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να το προτείνουμε. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ επίσης αναφέρθηκε σε πολύ συγκεκριμένα θέματα και επίσης η δημιουργία ενός ταμείου το οποίο θα καταστήσει με πραγματικούς όρους αντιληπτεί την διαδικασία αυτή από το ευρωπαϊκό κοινό. Δεν είναι τόσο απλό βέβαια το θέμα. Δεν αρκεί να πούμε ότι κοιτάξτε το βασικό είναι να συμφωνήσουμε στην πρώτη ανάγνωση και από εκεί και πέρα θα δούμε. Δεν θα σας καθασταρίσω άλλο δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλες τις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσα σαν σκιώδης εισηγητής. Θα τις εξετάσετε και θα τις εξετάσουμε από κοινού με πνεύμα συνεργασίας. Και θα ομαδοποιήσουμε πάρα πολλές νομίζω μεταξύ τους τροπολογίες. Είναι βασική ευθύνη των εισηγητών να συνεχίσουμε τη συνεργασία όπως αυτή που είχαμε άλλωστε και στο παρελθόν έτσι ώστε η πρώτη ψηφοφορία να είναι θετική. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο μα να καταλήξουμε σε αποφάσει με υψηλή πλειοψηφία στο εσωτερικό τη επιτροπή μα. Και σε αυτή τη φάση να μην σκεφτόμαστε στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στην περαιτέρω φάση. Ευχαριστώ, Πίτερ Σκίνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Βόρτμαν Κόλ, κατάφερε να τα χαρακτηρίσω αυτά κατά τρόπο, τον οποίο βρήκα μάλλον ανεπιτυχή εγώ τουλάχιστον Εθνικό πώ δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Κύριο Βρετανό, Βρετανός, ο οποίο ακολουθεί και τη γραμμή της Επιτροπής και τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου Σαλίση. Δυστυχώς όμως ο ε, κ. Βορτμαν Κόλ δεν έχει διαβάσει εκθέσει. Γι' αυτό κατέληξε σε διασφαλμένα ε, αποτελέσματα. Προτείνουμε αλλαγέ ω προ τι δημοσιονομικέ ευθύνε, προσδιορισμού, ορισμού, συμμετοχή των εμπλεκομένων στο επίπεδο που θα πρέπει να είναι, στο κατάλληλο επίπεδο, φιλοδοξίε για τις αρχές, ε, παρότι διαφωνούμε ω προς το κατά πόσον θα έχουμε την διάθεσή μα τον χρόνο και το χρήμα που χρειάζεται. Έχουμε επεκτείνει επίση την κοινή συμβουλευτική επιτροπή έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει τι αποφάσει τη σε πιο ισορροπημένο τρόπο και να μπορεί να προχωρεί Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ του δικού μας κειμένου και του κειμένου του Συμβουλίου. Δηλαδή, λίγο πολύ έχουμε προσθέσει νέα στοιχεία στο κείμενο της Επιτροπής τελευταία ώρα. το κείμενο είναι του Κοινοβουλίου και πρέπει εμείς να προσδορίσουμε την, ε, τις προτιμήσεις μας στην πραγματικότητα, το ρεαλισμό, τη λογική που θέλουμε. Μην μας πείτε ότι δεν είναι η ώρα τώρα να πούμε πώς θέλουμε να διαμορφωθεί το σύστημα με το οποίο θα δίνετε χρήματα μέσα από το Ταμείο τα επόμενα 6, τους επομενους 6-7 μήνες, καλό θα είναι να μπορούμε να τα καταφέρουμε μέχρι το Γενάρη ή αλλιώ θα πρέπει το πολιτικό μας κεφάλαιο να το εξαντλήσουμε προκειμένου να συστήσουμε ότι αποτύχαμε κυρία Καρσία Μαργκάιο στην προσπάθεια να συστήσουμε το συμβόλαιο αυτά που πρέπει να επιτύχουμε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εξαντληθούμε μόνο σε αυτά. Μπορεί να διαφωνούμε σε αυτά, σε ορισμένα σημεία του περιεχομένου, αλλά υπάρχουν σημεία στα οποία συμφωνούμε και εκεί πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες. Ας μην ε, σκεμαχούμε λοιπόν με το 5% του ΑΕΠ για ένα ταμείο στην 1η Ιανουαρίου που ε, θα πήγαινε τις δικές σας, τις, ε, τους δικούς σας υπολογισμούς στο 55% επί του ΑΕΠ για τις τάξεις κλπ. Προφανώς είναι όλα λάθος, έτσι δεν είναι. Ε, βλέπετε δεν συμφωνήσουν όλοι. Ούτε και το ενεργητικό που θα χρησιμοποιούν ε, τα ταμεία. Μερικά έχουν να κάνουν με ε, συστήματα πλεονασματικά, τα οποία θα σημαίνουν ότι θα πρέπει στη Γερμανία και σε άλλα κράτη-μέλη να στήσουμε να αντιδράσουμε με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν διαφορετικέ λύσει λοιπόν, αλλά το θέμα είναι θέλουμε να χάσουμε χρόνο συζητώντα πράγματα με το Συμβούλιο έστω και χωρίς επιτυχ... επιτυχίας. Εγώ θα να κοιτάξουμε εκεί που μπορούμε να κερδίσουμε. υπάρχει το ζήτημα της, του κινδύνου της απώλειας του ηθικού πασκύρους. Γι' αυτό ίσως θα ήταν καλό και η Ελίσσα Φερέρας να κοιτάξει. Ναι, γιατί είστε κυρία Γκαρσία Μαρκαγιο πολύ γοητευτικός και μπορεί να την πείσετε, αλλά κάποια επιχείρηματα από τα δικά σας τουλάχιστον, εμένα δεν με πείσανε. Σιλβί, για να δούμε ποιος αντέχει. Θα είμαι πολύ σύντομη αφού μας ακούει τρεις κούκος εδώ μέσα. Ευχαριστώ αυτούς που έμειναν πάντως. Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο. Θέλουμε να προχωρήσουμε το χύτερο δυνατό. Δεύτερον, δεν θέλουμε να νερώσουμε το κείμενο. Είναι ουσιοδέστατη σημασία σε αυτό. Και συμφωνώ με τον Χωσέ Μανουέλ. Δεν θεωρώ ότι η συναπόφαση σημαίνει το απόφαση. Το, το Συμβούλιο ορίζει την τοποθεσία και το Κοινοβούλιο μετατοπίζεται πηγαίνει εκεί που θέλει το Συμβούλιο. Δηλαδή, όχι, θα κάνουν μια προσπάθεια και από τι δύο πλευρέ. Γιατί πολλέ φορέ έχουν ε, καταστραφεί κείμενα από τι εσωτερικέ αυτέ λογικέ του Συμβουλίου. Εγώ είμαι δεκτική σε κάθε πρόταση τροπολογία, σε κάθε πρόταση του Συμβουλίου που θα εξυπηρετούσε το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον, που θα εξυπηρετούσε το γενικό συμφέρον του στόχου που επιδιώκουμε. Δηλαδή, ενό πιο αποτελεσματικού συστήματο. Αν είναι έτσι, να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Αλλά εάν πει το Συμβούλιο, εγώ έχω ένα εθνικό όραμα, δείτε το και μέχρι εκεί πάω, δεν ξέρετε το ξεπερνώ, δεν ε, μπορώ να σας ακολουθήσω. Για δε τα ισπανικά μου δεν μπορώ να σχολιάσω περισσότερο, γιατί μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Για την κυρία Λούλιν και τον κύριο Πόρτος που έχουν φύγει, βεβαίω θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών και ανοίγματο υπάρχουν διαφορετικέ ευαισθησίε από ό,τι βλέπουμε, αλλά θα τη βρούμε την ισορροπία πιστεύω και με τον Πίτερ Σκίνερ θα συμφωνήσω πιστεύω. Έχουμε συνεργαστεί όλοι μαζί, θα συνεχίσουμε. Στην Επιτροπή Plus ίσως να υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία διαφωνούμε περισσότερο, αλλά θα τα βρούμε, θα τη βρούμε την άκρη. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μα περισσεύουν και 15 λεπτά. Θέλει κανεί να ξαναλάβει το λόγο. Όχι, τι κρίμα. Ευχαριστώ. Α κηρύξω το πέραστη συνεδριάσεω, συνεδριάσεως, απαλλάσσοντάς σας από περαιτέρω λεπτομέρειες αυτής της συζήτησης. Χαίρετε.